Ja, schönen guten Morgen. Liebe Kollegen. Καλημέρα σα, κυρίε και κύριοι, αξιότιμε κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχά, οι αποφάσει τη χθεσινή συνεδρίαση των συντονιστών. Σα τα αποστήλαμε όλα αυτά και αν δεν έχετε αντιρρήσει τι οποίε και να εκφράσετε μέχρι σήμερα το μεσημέρι, ε, θα θεωρήσουμε ότι είναι εγκεκριμένα τα πρακτικά Ύστερα, θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ στην αίθουσα μια ομάδα επισκεπτών της European Passengers Federation της Lucy Anderson. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιβατών. Να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Κατάρχά να ψηφίσουμε για την ημερήσια διάταξη. Αποφασίσαμε λοιπόν χθε ότι σήμερα πρόκειται να γίνει ψηφοφορία για το κατά πόσον θα αλλάξουμε ένα σημείο τη ημερήσια διάταξη. Υπάρχει λοιπόν ένα αίτημα να αλλάξει το 11, να διαγραφεί από την ημερήσια διάταξη. Ποιο είναι υπέρ τη διαγραφή παρακαλώ. Ποιο είναι κατά τη διαγραφή. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πώς είναι, ποιος είναι, μάλλον, έναξη ψηφοφορίας. Α, ένας υπεράριθμος από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, παρακαλώ. Για κοιτάξτε το. Εξακολουθεί να είναι ένας υπεράριθμος. Okay. Also die Abstimmung ist eröffnet. Wir stimmen ab über den Tagesordnungspunkt 11 zu Ψηφίζουμε λοιπόν για την διαγραφή του σημείου 11. Όπως είναι υπέρ, ψηφίζει... Όποιος είναι υπέρ της διαγραφής να ψηφίσει ναι, όποιος είναι κατά της διαγραφής να ψηφίσει όχι. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, τις άκουσα τις διαμαρτυρίες. πέρας 24 υπέρ, 22 κατά Διαγράφεται, διαγράφεται λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριο Αρτούγα, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το ότι έγινε αυτή η διαγραφή. Δεν υπήρχε συγκεκριμένο επιχείρημα για να διαγραφεί το συγκεκριμένο ψήφισμα. Πρώτη φορά σε 3,5 χρόνια εμφανίστηκε και πρότεινα οποιαδήποτε δυνατότητα και θα ήμουν διτεθειμένο να επεξεργαστούμε και ένα νέο κείμενο με του συναδέλφου. Άρα δεν ήταν αυτό τελικά δυνατόν. Και το δηλώνω ξεκάθαρα ότι αν έτσι εργαστούμε στο μέλλον, εγώ πραγματικά δεν είμαι διόλου σύμφωνο και αυτό θέλω να μπει και στα πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ, Λίγο Πρόεδρο. Το καταγράψαμε και περνάμε στι περαιτέρω ψηφοφορίε. Καταρχάς, λοιπόν, ε, η βιώσιμη κινητικότητα. Η Καρή Μαντέλη είναι η συγκεντρία. Τροπολογία 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78. Α, καταπίπτει. 82 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 6. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Amendment 88. 88 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος Συμβαστική 2 Υπέρ Κατά Αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 3 τώρα Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 160 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ένβη 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 151 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5α υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 143. 243. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 292. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 211 υπέρ κατά άποχες. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Η 211. Abstimmung ist eröffnet. Έναρξη. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. Αλλά πάλι υπεράριθμος ένας από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ναι, τώρα καλύτερα τα πράγματα. Έναρξη ψηφορίας παρακαλώ για την 211. Πέρα. 24 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. Σε μεβαστική 9. Υπέρ. Κατά. άποχέ, εγκρίνεται. Kompromiss 10. Wer ist dafür? 10 υπέρ. Κατά. Άποχε, εγκρίνεται. 209 4 9 Υπέρ. Κατά. Ας τα ελέγξουμε παρακαλώ. 203-4-5-6-7-8-9. Έναξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Παύλη. Πέρας. 26 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. Das folgt, jetzt kommt Kompromiss 11. Wer ist dafür? Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 225 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέντι 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, δεν είμαι σίγουρος. Ας το ελέγξουμε. Μου φαίνεται ότι απορρίπτεται. Ρέντζι 7. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρα. 20 υπέρ, 25 κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 81. Έναρξη ψηφορίας. Πέρασε. 19 υπέρ, 27 κατά απορρίπτεται. 245 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε πάλι παρακαλώ. παρακαλώ. ψηφοφορίας. Πέρας. 20 υπέρ, 27 κατά απορρίπτεται. Παράγραφος, συμβαστική 13 μάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 244 και 240. Υπέρ. Και 291. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ζητείτε έλεγχο για την ΕΔΙ 3. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορία. Πέρας. 24 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. Ρέτζι 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. NV4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ για την NB4. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρα. 20 υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτεται. 261 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε αυτή την τροπολογία, την 261 παρακαλώ. Έναρξη. Πέρας. 15 υπέρ 31 κατά απορρίπτεται. Η συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 224 ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 277 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 469 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας. 20 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. 361 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 478 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 287 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ για την 287 ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη. Πέρας. 20 υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται. Ρέτζι, 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 311. Υπέρ. Η συμβιβαστική 19. Συγγνώμη. Η συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα η 311 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε για να είμαστε σίγουροι. Για την 311 παρακαλώ έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 20 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. Η 464 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 433 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Η 349 υπέρ. Κατά. Α, ας το ελέγξουμε, ας το ελέγξουμε. Για την 349 παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος. 20 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. 327 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η ε, 358 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Η 358, η 358. Υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Η 363. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 389. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 360. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 387. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 454. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 391. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 392. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος συζητείτε για την 392. Πέρας. 20 υπέρ, 25 κατά απορρίπτεται. 393 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 3, 96, 97, 98, 99, 400, 401, 402. Υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 404. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 403. Καταπίπτει. Και η επόμενη. 407 ε, λοιπόν. Καταπίπτει και αυτή. Ένβη 11. Σε δύο τμήματα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται nb 2 δεύτερο τμήμα μάλλον της nb 11 υπέρ. Δεύτερο τμήμα υπέρ, παρακαλώ. Κατά. 411 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 429 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 434 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. το Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωται. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τετρακόσια υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ένα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 430 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 431 υπέρ αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 395 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 499 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 453 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 310 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 213 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Ρέτη 13 υπέρ. Κατά Αποχέ εγκρίνεται. Ρέτζι 9 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 14 ναι, υπέρ. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 459 460 461 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 461 ελέγχουμε την 461 παρακαλώ ηλεκτρονικά 23 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. Τετρακόσια υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 463 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 466 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η 467 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει συμβιβαστική 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική... Α, όχι, η 473 λέει ο πρόεδρος υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 501. Όχι, εντάξει, ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 473. 473 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρασε. 19 υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται. 501 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 326. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 388. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 489, 490, 491. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. 491. Πέρας. 16 υπέρ, 29 κατά απορρίπτεται. 492 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 494 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κατά πίπτη 493 και 95 ρέτζι 20 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές Ν2-8 NV8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γιατί 18. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν. Πέρας. 19 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. NV, α. Υπέρ. Κατά. Άποχες, εγκρίνεται. NVP, ρο, ελληνικό και η τροπολογία 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. NVQ και η 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε. Για την 30 παρακαλώ. ενάξει ψηφοφορία. Πέρας. 19 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 35, συμβαστική 35, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 19, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε προφορική τροπολογία, ο μικρόν α, oral amendment, της εισηγήτριας. Η κυρία Ντέλη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Αυτή η προφορική τροπολογία καταδεικνύει ότι η χρήση του δίζελ ε, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πιο φθηνό αυτό το καύσιμο γιατί δεν υπάγεται σε τόσο υψηλή φορολογία. Και μάλιστα για να δελεάσουμε τους καταναλωτές πολύ συχνά παρουσιάσαμε το πετρέλαιο κίνηση στο δίζελ ως πιο καθαρό, πιο φιλοπεριβαλλοντικό καύσιμο από τη βενζίνη. Αλλά στηριχθήκαμε σε ψέματα όλα αυτά τα χρόνια γιατί δίζελ καθαρό δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ένα ψέμα που έχει οδηγήσει σε πάνω από 400.000 προώρους θανάτου στην Ευρώπη το χρόνο. Οπότε δεν έχει λόγο αυτή η φορολογική ελάφρυνση του ντίζελ. Είναι αντίθετα απειλή στη δημόσια υγεία των Ευρωπαίων. Γι' αυτό σα καλώ να υπερψηφίσετε αυτή την ε, τροπολογία για να κοιτάξουμε επιτέλου κατάματα την πραγματικότητα. Να δοθεί ένα τέμα σε αυτή την άδεια για ρήπαση. Να καταργήσουμε το ντίζελ και να ενθαρρύνουμε τι πόλει και τα κράτη να περάσουν στη χρήση άλλη εναλλακτική, άλλου εναλλακτικού καυσίμου. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου, δυστυχώς, τα υπόλοιπα σχόλια της κυρίας Δελή. Μίκρο; Δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχουν αντιστάσεις κατά της προφορικής τροπολογίας αυτής. Θα πρέπει να σηκωθείτε όρθιοι. Αν είσαστε κατά της προφορικής τροπολογίας, παρακαλώ, θα πρέπει να σηκωθείτε. Και εφόσον είσαστε παραπάνω από τρεις, απορρίπτει την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα. Ψηφίζουμε λοιπόν την NVF Υπέρ. Κάτα. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. NVG. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Age ήτα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. NVI, γιώτα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. NVJ, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 48, υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. NVE. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Τροπολογία 32 καταπίπτει. Η 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 59. Έναρξη ψηφοφορίας. Δεν αριθμός έλκα αυτή τη φορά. ψηφοφορία, πέρα ψηφοφορία. Η 21 υπέρ, 26 κατά Η 60 υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Συμβουλή 37 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 38 υπέρ συμβαστική. Κατά. άποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στροπολογία 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. NV10. NVC υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Ένωση και κάπα υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. ελ υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. NVM ε μη υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Η 74 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ για την 74. Ένα ψηφοφορίας. Πάλι ένας υπεραριθμός από το ΕΛΚ όμως. Ωραία τώρα. Πέρασε. 20 υπέρ, 27 κατά απορρίπτεται. NVN, νη, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. NVO, Όμικρον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NVR. Ε, καταπίπτει. NVS υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ για την NVS. Ας γίνει η ηλεκτρονική συμφορία. Έναρξη. εγκρίνεται. NVT, ταφ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 δεν ψηφίζεται. Η τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 80. Α, δεν ψηφίζονται λοιπόν οι επόμενε τροπολογίε. Τελική ψηφοφορία λοιπόν. Ένταξη ψηφοφορία. Πέρασε. 37 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά και 5 εποχές. Η Καρή Μαντέλη, λοιπόν, εγκρίνεται η έκθεση και το λόγο έχει η κυρία Ντέλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επ' ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές μου, γιατί ήταν δύσκολο το έργο μας ε, της εκπόνησης συμβαστικών τροπολογιών. Τα καταφέραμε όμως και τους ευχαριστώ θερμά. Επίσης, ε, να ευχαριστήσω και τον Μινί Κρισμάκερ, ε, τον Πολ Μπέρκμαν, τον συνεργάτη μας για το καταπληκτικό του έργο και επίσης τη Μάγκη, τον Εμμανουέλ, τον Ματιέ, την Κιωμίν, που ήταν οι αφανείς ήρωες στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Τους ευχαριστώ όλους θερμά. Und Σας ευχαριστώ και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Η Μέρια Κιλόνεν είναι η εισηγήτρια. So, darf ich um Σας παρακαλώ, ησυχία. So, Kompromiss 1. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορριβέται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Δεύτερο τμήμα. Κατά μάλλον. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Κατά. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ για τη 12 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Geschlossen. 23. Πέρας. 23 υπέρ. 23 κατά ισοψηφία απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ή 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ τα 47. Την 44, συγγνώμη, το 44. Πέρα. 25 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 74. Ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφορίας. Πέρασε. 20 υπέρ, 25 κατά απορρέπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε και την 77 παρακαλώ. Ένα ψηφορίας. Πέρασε. 21 ψήφοι υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 85 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 41 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Με Μεριά Κίλεν, συγχαρητήρια. Και σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στις τρεις ψηφοφορίες για τα αποτελέσματα του τριμερού διαλόγου για το τεχνικό πυλώνα της δεσμής μέτρων για τους σιδηροδρόμους έχουν ήδη αποφασιστεί, αλλά πρέπει και επίσημα να ψηφιστούν. Και έτσι λοιπόν, καταρχάς την πρόταση του Βιλμπά Μπαραντίκα. Υπέρ. Ένταξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Ηλεκτρονικά θα γίνει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 38 η ψήφη υπέρ 4 κατά 3 Και τώρα περνάμε στην δεύτερη έκθεση. Κράμερο εισηγητής. Δεν τον ξέρω, λέει ο πρόεδρος. Έχουμε λοιπόν ε, ε, την ψηφοφορία. Πέρασε. 37 37η υπέρ, 5 κατά, 3 εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τρίτη ψηφοφορία, Ρόμπερτ Ζήλερ, ο οποίο ε, είναι στο τηλέφωνο. Α, δεν πειράζει, θα ακούσει το Πάει. Ένα ψηφοφορία. Πέρα. 38 υπέρ, 4 κατά, 3 αποχές, εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ και τους τρεις you. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 12. Και περνάμε στο 12 της μεταξύ από την Γενική Διεύθυνση ε, των αποτελεσμάτων του έλεγχου REFIT. Ένα σύντομο, σύντομο, σύντομο διάλειμμα ενός λεπτού για να εξέλθουν τι αιθούσε όσοι το επιθυμούν. Marek, this is Dominic's point now. Yeah. Okay, thanks. well done. Well done, Jehovah. Yeah.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 So, wir kommen jetzt zu Punkt 12. Θα περάσουμε τώρα στο 12. Παρουσίαση από την Γενική Διεύθυνση μου για τη ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ασφάλειας των επιβατικών πλοίων. Λάβαμε τα αποτελέσματα του ελέγχου REFIT ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ε, τα πρότυπα ασφάλειας. Από το έγγραφο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνουμε ότι η νομοθεσία γραμμέ εκπληρώνει του στόχου του. Αλλά σε γενικέ γραμμέ επίση σκεφτόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει και μια απλούστευση τη οδηγία. Έχουμε δύο νομοθετήματα τα οποία επικαλύπτονται και αυτό θα πρέπει να επιληθεί για να ε, ενισχυθούν τα πρότυπα ασφαλείας. Και έχουμε λοιπόν υπόψη και το Κονκόρδια και το Φλαμίνια και έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει μια πρωτοβουλία για την απλοποίηση και τη βελτίωση τη σχετική νομοθεσία για τα επιβατικά πλοία. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση ε, MOVE για να μας παρουσιάσει εκτενώς τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ριφίτ, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, για την, ε, στην ατζέντα προβλέπετε αυτό. Ε, προβλέπετε αυτό για πιο μετά. Είναι δίκιο έχετε λίγο ο Πρόεδρος, άμα δεν είναι η Επιτροπή, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι 10 και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

Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, συνεχίζουμε. Είναι 10 και 4 ακριβώς και συμφωνούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, παρακαλώ καθίστε. Αν δεν θέλετε να παρακολουθήσετε τη συνέχεια της συνεδρίασης, παρακαλώ βγείτε έξω από την αίθουσα. Η εισαγωγή έχει ήδη γίνει, οπότε να δώσω το λόγο κατευθείαν στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη με την παρουσίασή μου για να γίνει η συζήτηση μετά. Να εξηγήσω όμως σήμερα στην Επιτροπή πώς επανεξετάσαμε στο λεγόμενο fitness check την αρακή νομοθεσία που εφαρμόζεται για τα επιβατικά πλοία. Εδώ και δύο χρόνια περίπου, διότι πρόκειται για μια περιοχή αρκετά τεχνικής και περίπλοκης φύσεως με διάφορα επίπεδα νομοθεσίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών ναυτιλίας. Μεγάλα τμήματα της νομοθεσίας έχουν, που είναι εφαρμόσιμα έχουν δημιουργηθεί στα, στα 15 τελευταία έτα, έτη, με συγχωρείτε, και αυτό για να ανταποκριθούμε σε ατυχήματα που είχαν συμβεί. Έχουμε τέσσερις βασικές δέσμες νομοθεσίας. Τεχνικές προϋποθέσεις των σκαφών σε εγχώριες μετακινήσεις, επιθεωρήσεις και έλεγχοι που εφαρμόζονται, συγκεκριμένη νομοθεσία κατόπιν του ναυαγίου του Εστόνια για τα ρόπαξ φέρεις και επίσης για την καταχώρηση των επιβατών άλλη μια δέσμη. Έχουμε εξετάσει λοιπόν πώς συνδυάζονται όλες αυτές οι ιδέες με τις νομοθεσίες και πώς μπορούμε να τις βελτιώσουμε. Τώρα ένα πλαίσιο για να εξηγήσω για ποιο λόγο αυτό είναι σημαντικό και ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε περίπου 400 εκατομμύρια επιβάτες το έτος που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται από τα σκάφη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμένων έχουμε 210 περίπου εκατομμύρια επιβάτες που μεταφέρονται μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμένων και στις εγχώριες μετακινήσεις σε περίπου 120 εκατομμύρια, δηλαδή επιβάτες που μετακινούνται εντός λιμένος, λιμένων του αυτού κράτους μέλους και για να διευκρινίσω κάποιους ορισμούς σχετικά με το τι είναι επιβατικό σκάφος και πώς το διακρίνουμε από γιότ ή κρουαζιερόπλιο. Πρόκειται για σκάφος μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες που η δαλος είναι σκάφος αναψυχής και τα σκάφη αναψυχής διέπονται από άλλη οδηγία, την οδηγία για τα σκάφη αναψυχής και ίσως κάποιοι από εσάς να έχουν οδηγήσει και κάποιο τέτοιο. Τώρα, τα ευρωπαϊκά σκάφη μπορεί να είναι φέρι και υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία των φέρει που υπό την έννοια της ασφάλειας είναι πολύ σημαντικά είναι τα ρο-ρο ή ροπαξ στα οποία που επιβιβάζεται κανείς μαζί με το αυτοκίνητό του και μπορεί και να έχει καμπίνα διανυκτέρευσης και τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο ανατροπής σε περίπτωση ζημιάς στο κέλυφος του σκάφους διότι αν υπάρξει σοβαρό ατύχημα τα πράγματα κινούνται γρήγορα και γι' αυτό το 2003 υιοθετήθηκε νομοθεσία μετά το ναυάγιο του Εστόνια για ακριβώς αυτού του είδους τα σκάφη. Τώρα, τι ρυθμίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία οι σχετικέ διατάξεις των οδηγιών για την ναυπήγηση, την ασφάλεια σε πυρκαγιά, διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες μαζί με τον εξοπλισμό των σωσιβίων, της διάσωσης ε, και τα λοιπά. Έχουμε και τις ε, ούτως αποκαλούμενες επιθεωρήσεις ή τους ελέγχους σε βάση περιπτώσει ασφαλείας και την καταχώρηση των επιβατών. Και για να εξηγήσω κάπως την περιπλοκότητα των διαφορών επιπέδων, σκεφτείτε ένα σκάφος που κινείται μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Θα ήταν διεθνής μετακίνηση και επομένως θα ίσχυαν προϋποθέσεις IMO. Αν είναι φέρει ρόπαξ, πέραν των απαιτήσεων IMO θα υπήρχαν και ευρωπαϊκές και θα επανέλθω σε αυτό για να σας εξηγήσω γιατί. Διεθνής μετακίνηση θα ήταν και μετακίνηση μεταξύ κράτους μέλους και τρίτου κράτους, π.χ. από την Ελλάδα προς την βόρεια ακτή της Αφρικής, σε αντίθεση με εγχώριες μετακινήσεις που όπως σας έλεγα πριν δηλαδή μεταξύ λιμένων του αυτού κράτους μέλους, όπου εκεί δεν θα ίσχυαν οι υποθέσεις IMO, αλλά η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσπαθούν να ενσωματώσουν τις αυστηρές διεθνείς διατάξεις, οι οποίες συνήθως προβλέπουν μεγάλα σκάφη που κινούνται σε ανοιχτές θάλασσες και ωκεανούς και όχι σε πιο κλειστά νερά ας πούμε. Οι θαλάσσιες περιοχές που περιβάλλουν την Ευρώπη και οι συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες κινούνται τα σκάφη αυτά είναι αρκετά διαφορετικές και επομένως οι διατάξεις ασφαλείας εφόσον πρέπει να είναι ίδιες για όλα τα σκάφη ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι υπερβολικές ή αν ένα σκάφος έχει να πηγηθεί για πιο ρηχά ύδατα όπως τη Βαλτική δεν θα είναι κατάλληλο για να πλεύσει στις ε, δυτικές θάλασσες της Ιρλανδίας. Εξού και το υφιστάμενο καθεστώς προβλέπει εξαιρέσεις για τα κράτη-μέλη οι οποίες εξαιρέσει θα πρέπει να ελέγχονται από την ε, Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ε, Ασφάλεια Θάλασσα. Και συνοψίζοντας στην επόμενη διαφάνεια, η νομοθεσία μας καλύπτει σκάφη των εγχωρίων αυτών μετακινήσεων και των διεθνών διατάξεων για τα ferry ΡΟΠΑΞ και τις ε, προϋποθέσεις καταχώρησης. Ε, ήμουν τον Ιανουάριο εδώ με τον κύριο Καραμίτσο μετά από το κρούσμα στο Βόρειο Ατλαντικό με σκάφος που υπέστη πυρκαγιά σε μετακίνηση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας πρόκειται πρόκειτο για διεθνή μετακίνηση όπου ίσχυαν και οι ευρωπαϊκές διατάξεις θα επανέλθω σε αυτό στα πορίσματά μας διότι θεωρούμε ότι εκεί κάτι πρέπει να αλλάξει. Τώρα, πρέπει να προσέξουμε το εξής. Εδώ μιλούμε για προϋποθέσεις για σκάφη εγχωρίων μετακινήσεων τα οποία δεν θα ίσχυαν για την περίπτωση σκάφους όπως το Κώστα Κονκόρντια, κρουαζιερόπλιο δηλαδή, το οποίο δεν φέρει σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο κινείται στη Διεθνή θάλασσες. Στην Καραϊπική, στην Ασία και επομένως οι προϋποθέσεις για το σκάφος και το πλήρωμά του πρέπει να υπόκεινται στους διεθνείς οργανισμούς προς τους οποίους εμείς πρέπει να παρέχουμε input για να βελτιώνονται οι διατάξεις αυτές διατηρώντα υπόψη είναι ότι έχουμε περί τα 6 εκατομμύρια Ευρωπαίου κάθε έτο που μετακινούνται με τέτοια γεροπλήγα και οι οποίοι οι πολίτε δεν επιλέγουν τα σκάφη ανάλογα με τη σημαία. Τώρα, γιατί ρυθμίζουμε τα επιβατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι τα διεθνή πρότυπα είναι επαρκή. Η απάντηση είναι ότι πρώτον, τα διεθνή πρότυπα δεν ισχύουν στα εγχώρια ύδατα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα καθεστώς ασφαλείας και ένα καθεστώς για την εσωτερική αγορά που να ισχύει για τα εγχώρια ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κράτη-μέλη. Και βεβαίως θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει και σε επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από καταστροφικά ατυχήματα που είχαμε ιδιαίτερα με τάνκερ, με δεξαμενόπλια και σκέφτομαι εδώ το Prestige για παράδειγμα έχουμε τον οργανισμό για την ασφάλεια στη θάλασσα επί τη βάση διεθνών διατάξεων και προτύπων αλλά έχουμε δημιουργήσει το αυστηρότερο πλαίσιο ασφαλείας για τις θαλάσσιες μετακινήσεις στον κόσμο. Ο οργανισμός επισκέπτεται όλα τα κράτη-μέλη και ελέγχει την υλοποίηση, την εφαρμογή της νομοθεσίας, το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση των διεθνών οργανισμών. Και σε περίπτωση παραβιάσεων οδηγούνται οι παραβάτες, τα κράτη-μέλη, στο δικαστήριο. με τα διεθνή πρότυπα θα ήταν δύσκολο να έχουμε κοινό επίπεδο προτύπων και για την εσωτερική αγορά. Τραπορίσματα είναι κατάλληλη η ορακή νομοθεσία για τους στόχους που έχει θέσει και εδώ προσπαθούμε να προσμετρήσουμε διάφορα ατυχήματα και τη διάσταση της εσωτερικής αγοράς. Καταρχάς, να σας δώσω μια εικόνα για πόσα σκάφη μιλούμε. Έχουμε 922 επιβατηγά αυτή τη στιγμή σε εγχώρια ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιημένα υπό την οδηγία Δηλαδή το 1 τρίτο περίπου του συνόλου των επιβατικών σκαφών. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός είναι μικρός αριθμός. Γιατί αν τον συγκρίνει με σκάφη ξύλινα ή συνθετικά, διότι η οδηγία μας ισχύει μόνο για μεταλλικά σκάφη, θα έλεγε κανείς ναι, είναι μικρός αριθμός. Αν όμως λάβει υπόψη του κανείς τον αριθμό των επιβατών, είναι σαφές ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει περί τα δύο τρίτα του συνόλου της δυνατότητας μεταφοράς επιβατών. Που είναι λογικό. Γιατί όσο πιο μεγάλο είναι το σκάφος, τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση να, να φυγείται από χάλιβα και επομένως μεγαλύτερη δυνατότητα μεταφοράς επιβατών. Περί τα δύο τρίτα λοιπόν των σκαφών που εμπίπτουν στη δυνατότητα μεταφοράς επιβατών δηλαδή 380 χιλιάδες εμπίπτουν στην νομοθεσία. Νομοθεσία που, όπως έλεγα, εφαρμόζεται για μεταλλικά, χαλίβδινα ή αντίστοιχα σκάφη. Και εδώ πάμε στο πρώτο θέμα που έχουμε εντοπίσει. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα έπρεπε να εφαρμόζεται και για το χάλιβα και για αντίστοιχα υλικά δεν είναι σαφές σε διάφορα κράτη-μέλη αν σκάφη ε, ναυπηγημένα από αλουμίνιο που είναι μέταλλο αλλά δεν έχει την ίδια αντοχή στην πυρκαγιά μπορεί βεβαίως να προστατευτεί να μονοθεί θα ενέπιπτε ή όχι στις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και προκειμένου να έχουμε ισότιμο παιχνίδι ίσους κανόνες για όλους το πόρισμα είναι ότι πρέπει να διαφαινιστεί αυτό. Επίση πρέπει να διαφενιστεί κατά πόσον τα σκάφη που εμπίπτουν στην οδηγία είναι σκάφη που κινούνται εκτός των λιμένων. Μπορεί κάποιο να κλείσει ένα ταξίδι από το λιμάνι του Αμβούργου για να κάνει έναν περίπλου το οποίο δεν θα ενέπιπτε το σκάφος αυτό δεν θα είναι έπιπτε στην νομοθεσία των σκαφών που βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα. Έχουμε δει ότι μόνον 70 μικρά σκάφη αυτή τη στιγμή κάτω των 24 μέτρων εμπίπτουν στην οδηγία, ενώ έχουμε σχεδόν 2.000 επιβατικά που δεν έχουν πιστοποιηθεί υπό την οδηγία. Και εδώ έχουμε ένα θέμα αναλογικότητας. Αυτά τα 1880 μη πιστοποιημένα σκάφη είναι μικρά, κάτω των 24 μέτρων, από συνθετικά υλικά και είναι σαφές ότι οι υφιστάμενες διατάξεις δεν είναι κατάλληλες για την αφήγηση αυτών των σκαφών. Χρειαζόμαστε λοιπόν άλλα πλαίσια κανόνων διατάξεων και για να είμαστε αναλογικοί για αυτά τα μικρά σκάφη για τα οποία έχουμε βρει ότι δεν υπάρχει εσωτερική αγορά φτάσαμε στο πόρισμα ότι δεν θα έπρεπε να καλύπτουμε υπό την, οδηγία, υπό την οδηγία αυτή σκάφη μικρότερα των 24 μέτρων. Τώρα, τι διαβουλεύσεις κάναμε στα πλαίσια της άσκησης αυτής. Είχαμε άμεσες επαφές με τις εθνικές αρχές και τους οργανισμούς για τις θαλάσσιες μεταφορές για να συλλέξουμε την εμπειρία των 15 ετών της εφαρμογής των διατάξεων αυτών. Κοιτάξαμε την περιπλοκότητα του ρυθμιστικού πλαισίου για να δούμε πώς μπορούμε να απλουστεύσουμε επιτρέποντας βεβαίως το ίδιο επίπεδο ασφαλείας και στην ιστορική αγορά προσπαθήσαμε να καθορίσουμε πώς τεχνολογικές εξελίξεις πρόοδος που έχει σημειωθεί στα τελευταία 15 χρόνια μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα. Κοιτάξαμε τι έχει συμβεί σε διεθνές επίπεδο και τι διδάγματα έχουμε από τα σημαντικά ατυχήματα που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Και το λέω ανοιχτά, προσπαθήσαμε να έχουμε ένα διάλογο των ενδιαφέρων μερών που είχαμε με τη βιομηχανία και με τις αρχές, αλλά ήταν δύσκολο να τον έχουμε αυτόν με τις ενώσεις των επιβατών. Διότι μία από τις αδυναμίες που έχουμε σε αυτό τον τομέα είναι ότι δεν έχουμε σχεδόν ενώσεις που θα προστάτευαν τα συμφέροντα των επιβατών. Για το μέλλον λοιπόν θα πρέπει να σκεπτούμε μαζί και εδώ υπολογίζουμε στη βοήθεια του Κοινοβουλίου πώς να ενισχύσουμε το διάλογο με ενώσεις επιβατών ώστε να είναι και η δική τους φωνή ισχυρή τη στιγμή που επεξεργαζόμαστε διατάξεις ασφαλείας επιβατών. Τώρα σχετικά με τα ατυχήματα και προκειμένου να αξιολογήσει κανείς κατά πόσον είναι επαρκής η υφιστάμενη νομοθεσία. Εξετάσαμε την τράπεζα δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για σχετικά με τα ατυχήματα και υπό την οδηγία από το 2009 για την έρευνα των ατυχημάτων έχουμε καθορίσει 408 ατυχήματα πιστοποιημένων σκαφών που μπορεί να φαίνεται υψηλός αριθμός αλλά τα περισσότερα από αυτά ήταν ατυχήματα χωρίς θύματα και χωρίς σημαντικές ίσως ζημίες είχαμε μία απώλεια ζωής και συγκρίνοντας τα δεδομένα τα μέσον όρο αυτά τα σκάφη μάλλον συνολικά είχαμε δύο κατά μέσον όρων τραυματισμούς και μόνο μία απώλεια ζωής όπως σας έλεγα ανά 100 ατυχήματα. Αν αυτό το συγκρίνει με τα σκάφη που κινούνται συνολικά και τα σκάφη που δεν έχουν δηλαδή ευρωπαϊκή σημαία που κινούνται στα εγχωρία η κατάσταση είναι διαφορετική. Υπάρχει τραυματίας κάθε δύο ατυχήματα και μία απώλεια ζωής κάθε 27 ατυχήματα. Και βεβαίως η περίπτωση του Κώστα Κονκόρδια σήκωσε τα μαγεία αυτά, τα ανέβασε. Και για να σας δώσω μια συγκριτική ιδέα, εδώ έχουμε τον κίνδυνο αναώρα μετακίνησης του επιβάτη και σε σύγκριση με άλλες, ε, άλλους τομείς μεταφοράς η απόδοση είναι ακόμα πολύ καλή. Βεβαίως εδώ τα αεροσκάφη είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα καθότι κινούνται πολύ πιο γρήγορα και επομένως το ατύχημα ανά ώρα κατέρχεται. Εδώ μιλούμε για ατομικά επίσης δεδομένα. Αν τα συγκρίνει με τον εταιρικό κίνδυνο, το Α380 έχει 500, το αεροσκάφος έχει 525 επιβάτες, ενώ τα κρουζιερόπλαια έχουν 6.000 επιβάτες. Επομένως, όταν υπάρξει πολύ σοβαρό ατύχημα έχουμε τελείως διαφορετικά νούμερα από την πτώση ενός αεροσκάφους. Ένα από τα απορίσματα ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία οπωσδήποτε υποστήριξε προώθησε τις ε, πωλήσει σκαφών μεταξύ των κρατών μελών. Έχουμε περί τα 400% αύξηση των σκαφών με ευρωαϊκή σημαία Συνολικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι ακόμα κατάλληλη η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά μπορούμε να την απλωστεύσουμε και εδώ έρχομαι στις τελευταίες τρεις διαφάνειες, ποιες είναι οι δράσεις που προτείνει η Κομισιόν για το μέλλον. Πρώτον, βρήκαμε ότι υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ διαφόρων καθεστώτων επιθεώρησης. Έλεγχοι που είναι υποχρεωτική υπό την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ευρωπαϊκούς λιμένες και εδώ προσπαθούμε να διαλευκάνουμε λίγο το τοπίο για να είναι και σαφέστερο και για τους ε, υπευθύνου. και πρέπει κανείς να δει τις ε, εφαρμοστές διατάξεις για τα μεγάλα σκάφη να υπάρξει άρση των δυσανάλογων προϋποθέσεων για τα μικρά σκάφη 70 εκτός σε σύγκριση με 2.000 εντός να δούμε την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος για τα σκάφη εκεί που δεν εμπίπτουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα έπρεπε να έχουμε αντίστοιχες δηλαδή διατάξεις όπως και έχουμε και για τα σκάφη αναψυχής και να χρησιμοποιήσουμε τα υφιστάμενα συστήματα υποβολής ε, εκθέσεων σχετικά με τα μεγέθη, τους αριθμούς των επιβατών. Οπότε όταν έχουμε ατύχημα όπως το Norman Atlantic να έχουμε άμεσα τον κατάλογο των επιβατών και τον αριθμό, ανάλογα με το είδος του σκάφους και να μην χρειάζεται στα μέσα της νύχτας να καλέσουμε κάποιον υπεύθυνο τηλεφωνικής επικοινωνίας για να μας στείλει τον κατάλογο. Και καλό θα ήταν να συμπεριλαμβανόταν και η υπηκότητα των επιβατών γιατί δεν έχει έτσι ακόμα ως προς τις διατάξεις αλλά σε περίπτωση σημαντικού ατυχήματος είναι σημαντικό να μπορούμε να ερχόμαστε άμεσα σε επαφή με τα προξενία ή τις πρεσβείες καθότι έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες που δεν φέρουν αναγκαστικά ευρωπαϊκό διαβατήριο. Και ένα τελευταίο σχόλιο για το διεθνές επίπεδο θα πρέπει να παράσχουμε και το κάνουμε ήδη input στον IMO για την βελτίωση της σταθερότητας των ευρωπαϊκών σκαφών και για οποιαδήποτε ζημιά στο εξωτερικό κέλυφο του σκάφους προκειμένου να συζητηθεί στον IMO την ερχόμενη άνοιξη. Συγκεκριμένες λοιπόν προτάσεις για τον IMO και εσωτερικά ένα καθεστώς ένα καλύτερο καθεστώς υποβολής εκθέσεων για τα φέρει ρόπαξ και εφαρμοστεία πρότυπα, ιδιαίτερα για τα μικρότερα σκάφη. Είναι περίπλοκο το θέμα, προσπάθησα να είμαι όσο σύντομη και απλή μπορούσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς εκτός μικροφώνου. Δυστυχώ θα πρέπει να σα ασκήσω λίγο κριτική, όχι μόνο επειδή καθυστερήσατε, αλλά είχαμε συμφωνήσει 10 λεπτά και τώρα μιλήσατε 25 λεπτά. Και δεν έχουμε και μεγάλε ε, ε δυνατότητε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση τη ε, του χρονοδιαγράμματος. Σας παρακαλώ στο μέλλον να είμαστε λίγο πιο συνεπείς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Βίνκ που έχει το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κατανοώ την κριτική που ασκήσατε, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι η παρουσίαση ήταν εξαιρετική και σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για αυτήν. Όντως, ε, το θέμα ήταν ε, το χρονικό πλαίσιο, όχι το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο ήταν εξαιρετικό. Είναι λοιπόν ε, μεγάλος ο πειρασμός σε αυτές τις περιόδους ε, του refit και της καλύτερης νομοθεσίας, better regulation, να κοιτάξουμε και τις... Ε, Εγώ εδώ θέλω να επιστήσω ιδιαίτερη προσοχή. Ως πολιτικοί είμαστε οι πρώτοι που θα διαμαρτυρηθούν σε περίπτωση ενός δυστυχήματος. Αλλά αν μπορούμε να προλάβουμε ένα δυστύχημα με την ομόθεσία, κοιτάξτε πώς είμαστε στην αίθουσα. Απουσιάζουν λοιπόν, λάμπουν τις απουσίας τους οι πολιτικοί. Ελπίζω λοιπόν αυτό να μεταφερθεί και προς τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς να επιμείνει σε αυτό το ζήτημα της ασφάλειας στις μεταφορές αυτές. Κατά δεύτερον, είναι δύσκολη, θεωρώ, εξακολουθεί να είναι δύσκολη η σχέση μεταξύ IMO και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γιατί δεν μπορεί να υιοθετήσει ο IMO τι ίδιε ε, προδιαγραφέ ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι υψηλό το επίπεδο ασφάλειας το οποίο έχουμε. Αυτό ήταν το δεύτερο. Κατά τρίτον, δεν κατάνοω το, Κόνστα, το Κώστα Κονκόρδια. Όταν ε, περνά στα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά βγαίνει από τα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς είναι δυνατόν να μην ισχύουν πλέον οι προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν σωστά κατάλαβα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί συμβαίνει αυτό. Ένα, δεύτερο, ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι το θέμα του enforcement, της ε, εφαρμογής δεν άκουσα να το αναφέρετε αυτό. Ποιος το έχει αναλάβει και πώς. Κα, τέλος, ε, καταλάβαμε τι είπατε για τις οργανώσεις επιβατών και στους σιδηροδρόμους και στις οδικές μεταφορές θα αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό. Θα πρέπει να αφιερώσουμε πιο πολύ προσοχή. Το θέμα του καταναλωτή φυσικά είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ΙΜΚΟ, αλλά σίγουρα θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ja, schön, Dank. Äh. Ο κύριο Ερτούγκ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπέρκ, για την πάρα πολύ καλή αυτή παρουσίαση. Παραδειγματικά ποια είναι η κατάσταση. Το τι συμβαίνει το ξέραμε και αυτό ισχύει και για τις εσωτερικές πλήτες αλλά και για τα πλοία ανοιχτής θαλάσσης. Δεν θα ήθελα να αναφέρω την πλευρά του, των εργαζομένων. Ξέρουμε ότι είναι πολλές οι υπηκότητες που απασχολούνται και εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες που ισχύουν. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Το θέμα είναι όμως καταρχάς η ασφάλεια, η ασφάλεια των πλοίων. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Refit check, έλεγχος ε, refit για την καλύτερη νομοθεσία για την ασφάλεια των επιβατηγών πλέον. Ε, θα υποβάλλετε καινούρια νομοθεσία, κάποια ανακοίνωση. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα της μελέτης της οποίες και αναθέσατε και η οποία κατέληξε σε πολλά και ενδιαφέροντα απορίσματα. Και στα ατυχήματα και στα δυστυχήματα που προκλήθηκαν ε, υπήρξαν και θάνατοι θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και το Norman Atlantic και το Costa Concordia αποτελούν ξεχωριστέ ενότητε, αλλά δεν θέλουμε να παρουσιαστούν στο μέλλον και άλλα τέτοια δυστυχήματα. Ερωτώ λοιπόν, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον και πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στο μέλλον, ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, η Τζάκη Φώστερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πολύ περιεκτική της παρουσίαση. Μάλλον δίκιο έχετε που τα φύγετε όλα αυτά, αλλά κάτι που είπε ο συνάδελφος είναι ότι έχουμε ισχύουσα νομοθεσία. Και ποιος ο λόγος, ποιος ο, λόγος ύπαρξής της είναι η εφαρμογή. Και σίγουρα θα θέλαμε μεγαλύτερη διαφάνεια, ε, ιδιαίτερα στη διαλεύκανση δυστυχημάτων ή ναυαγίων. Εγώ θα ήμουν πιο επιφυλακτική πάντως, γιατί θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ κατάγομαι από ένα ε, κράτος με μεγάλη ναυτιλία και καλό θα είναι να γίνεται διάκριση μεταξύ των εθνικών ε, ε, κανόνων, των ευρωπαϊκών, του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού. Όταν έχουμε τόσο περίπλοκο πλέγμα κανόνων, δεν ξέρουμε τι να εφαρμόσουμε. Και Είμαστε και μέλη του ΜΟ. Και τι γίνεται, γιατί τα πλοία πολύ συχνά αλλάζουν δρομολόγια. Ποιοι κανόνες ισχύουν. ισχύουν. Θα πρέπει όλοι να εφαρμόσουν τους ίδιους κανόνες. Και θυμάμαι την ακρόση που είχαμε για το Έρικα. Φυσικά κάναμε ακρόση και για το Κώστα Κονκόρντια. Το θυμάστε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Και σίγουρα πολύ συχνά συμβαίνουν ατυχήματα και ναυάγια. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα τι επιδιώκεται. Γιατί λέτε ότι υπάρχει νομοθεσία, εντάξει, νομοθεσία υπάρχει. Λέτε ότι είναι κατάλληλη, πολύ ωραία. Πιστεύω ότι μετά τα προβλήματα που είχαμε και τα μεγάλα ναυάγια και δυστυχήματα που είχαμε με τα ferry boat υπάρχει βελτίωση. Αλλά ποιος είναι ο στόχος σας, τι επιδιώκετε. Μπορεί να φαίνομαι ανόητη, αλλά πραγματικά δεν κατάλαβα τι σκοπεύετε να κάνετε. Απλώς μας κάνετε μία παρήθμιση του ιστορικού, του υποβάθρου, εντάξει, αλλά δεν μας λέτε τι πρόκειται να κάνετε. Είπατε να πλουστεύσετε την νομοθεσία. Ποια ακριβώς ε, νομοθετικά μέτρα θέλετε να πλουστεύσετε. Και ποια είναι η γνώμη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τις προτάσεις σας. Ίσως θα πρέπει αυτό να διαρευνήσετε πρώτα μέχρι τον Ιανουάριο και μετά να μας πείτε τα σχόλια του IMO. Αυτά ε, εκ μέρους της ομάδας συντηρητικών και μεταρρυθμιστών προς το παρόν. Κυρία Μάισνερ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Μπέρκη για την παρουσίαση αυτή. Πήρε παραπάνω ώρα από ό,τι προβλεπόταν, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή και μας έδωσε μια καλή επισκόπηση. Αυτό που είναι λίγο κρίμα είναι ότι δεν ε, κοιτάξαμε το περίπτωση του Ισλαμίνια γιατί ήταν, ε, δεν ήταν επιβατικό πλοίο. Δεν αφορούσε ε, επιβάτες, αλλά και πάλι έπεσαν νεκροί. Ένα άλλο θέμα. Είπατε ότι στο Κώστα Κονκόρδια δεν ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες και νομοθεσία. Μα πώς γίνεται αυτό, άμα κινείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πάντα να ισχύουν ευρωπαϊκοί κανόνες. Ε, γιατί ισχύει κάτι τέτοιο λοιπόν. Στην αυτιλία ισχύει κάτι άλλο. Επίσης δεν κατάλαβα ε, ε αυτό που είπατε ότι στις εγχώρες εσωτερικές μεταφορές δεν ισχύουν οι κανόνες του διεθνούς του οργανισμού. Πώς γίνεται αυτό, εγώ υποθέτω ότι ισχύαν, υπέθεσα ότι ισχύαν πάντα οι κανόνες του IMO, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τα άλλα σημεία τα οποία αναφέρατε τώρα. Εγώ κατάλαβα ότι μας ε, είπατε τι προτίθεστε να κάνετε όπου υπάρχει αλληλεπικάλυψη στην νομοθεσία, να γίνει μια πλούστευση. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ καλό και σημαντικό αν υπάρχει διπλή ρύθμιση. Ύστερα, για τα πλοία τα οποία είναι κάτω από 24 μέτρα, αν θα ήταν καλό να μην ρυθμίζονται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια και κάνουν μόνο ε, εθνικέ ε, μεταφορέ και μήπω θα πρέπει να μείνει στα πλαίσια της επικουρικότητας αυτό το θέμα. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσον οι κανόνες ε, οι οποίοι ισχύουν θα εφαρμοστούν παντού εξίσου και κατά πόσον ως Ευρωπαίος πολίτης αν κάποιος βρίσκεται σε ένα ε, χώρο ταξίδι πραγματικά ε, έχει τις ε, σωστές προδιαγραφές. Ύστερα, για την καταχώρηση θα πρέπει όντως να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι σε περίπτωση δυστυχήματος. Και επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε τις διάφορες ε, ε, κατηγορίες ε, πλοίων. Να δούμε μήπως πρέπει να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη προδιαγραφή, γιατί ως Ευρωπαίοι πολιτικοί ασφαλώς θα πρέπει να φροντίσουμε το θέμα της ασφάλειας των μεταφορών για τους επιβάτες. Και αν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο αυστηροί από τους διεθνείς κανόνες, γιατί να μην κοιτάξουμε πιο πολύ και να μην προωθήσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κριστίν Μπέρκ, για την πολύ καλή της παρουσίαση. Πιστεύω ότι μπορούμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι η ασφάλεια των μεταφορών και η προστασία των επιβατών ε, είναι θεμελιώδους σημασίας. Και σίγουρα δεν αρκούν οι μέτρα σε αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει απλώς να περιοριζόμαστε στις ε, εξοικονομής χρημάτων, γιατί μπορεί μερικές φορές να κάνουμε οικονομίες, αλλά να έχουμε μεγάλες απώλειες ανθρώπινες ζωές. Επίσης, η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα ασφάλειας είναι πολύ σημαντική. Κανένα κράτος μέλος και κανένας πολιτικός ε, δεν θα ήθελε να είναι μάρτυρες σε ναυάγια ή να χρειάζεται να θρύνει θύματα. Και κανένας δεν θα επικαλυστεί την επικουρικότητα όταν έχουμε ναυάγια και μάλιστα σαν θανατηφόρα. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα αναλογιστούμε και η πολιτική και τα κράτη-μέλη. Και το ίδιο και τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει από κοινού, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσουμε μια επικαιροποιημένη γνώση της πραγματικότητας και στην Ευρώπη και στον κόσμο και να αξιολογήσουμε την ασφάλεια του συστήματός μας ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Με τις νέες τεχνολογίες μπορούμε να εξυγχρονίσουμε το εξοπλισμό μας και θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα και διακλαδικά. Θα πρέπει όλοι να συνεργαζόμαστε στενά και να μην αγκιστρωνόμαστε στην αρχή της επικουρικότητας, γιατί εδώ το ζητούμενο είναι η προστασία των ανθρώπινων ζώων. Και αν θέλουμε διαλειτουργικά συστήματα, θα πρέπει να επιτρέψουμε και να διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Και εδώ έχουμε μια καλή ευκαιρία να διαμορφώσουμε ένα σύστημα που θα εξυπηρετήσει όλη την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει κοινέ δράσεις. Και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ξεχάσουμε λίγο την προσφυλή αυτή αρχή της επικουρικότητας. Γιατί εδώ το ζητούμενο είναι η, αύξη, η ενίσχυση της ασφάλειας και η διάσωση ανθρώπινων ζώων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Μπέρκ για την παρουσίαση που μας έκανε. Περιμένω ανυπόμονα να την διαβάσω πιο διεξοδικά. Γιατί εγώ έχω αναλάβει την έκθεση για το θέμα αυτό. Γι' αυτό και περιμένω ανυπόμονα να εγγύψω στο θέμα πιο ενδελεχώς. Και χαίρομαι που ασχολείστε με το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχετε διαβουλεύσει εκτεταμένε και με ομάδες ε, ε, συμφερόντων επιβατών. Και χαίρομαι που προτεραιότητά σα είναι η απλοποίηση της νομοθεσία. γιατί σίγουρα απευχόμαστε την ύπαρξη επικαλύψεων. Και συμφωνώ με, την, ε, με τις ανησυχίες και τον προβληματισμό της Γκεζίν γιατί τα περισσότερα πλοία έχουν, ταξιδεύουν σε διεθνή ύδατα. Έχουμε και την ε, περίπτωση του Κώστα Κονκόρδια. Ένα τμήμα του δρομολογίου όμως γίνεται σε ευρωπαϊκά ύδατα. Και σε τέτοια περίπτωση, όταν πρόκειται για διεθνέ δρομολόγιο, δεν ισχύουν καθόλου οι ευρωπαϊκοί κανόνε, ακόμη και στο, στο τμήμα του δρομολογίου που γίνεται σε ευρωπαϊκά ύδατα. Δεν το καταλαβαίνω. Φαντάζομαι θα υπάρχει κάποια λογική πίσω από αυτό. Γιατί θέλουμε να υπερισχύουν οι δικές μας νομοθετικές ρυθμίσεις όταν κάποιες, κάποια δρομολόγια γίνονται σε δικά μας χωρικά ύδατα. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς τα διάφορα ναυάγια, τα ατυχήματα, τους λόγους που οδήγησαν σε ατυχήματα και να βεβαιωθούμε ότι στο μέτρο του δυνατού αντιμετωπίζουμε τα αίτια των ατυχημάτων και των αβαγίων στην προσπάθεια βελτίωσης ε, της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας της ομοθεσίας. Ευχαριστώ. Well, thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω και πάρα πολλά να πω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι για μία φορά προσπαθούν κάπως να απλουστεύσουν το σύστημα και να βγάλουν κάποια περιπλοκότητα. Και αυτή είναι η μοναδική μου επιθυμία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είμαστε απλούστεροι και ακριβέστεροι όσο μπορούμε. Άρα δεν έχω κάποια αντίρρηση. Danke sehr. Jetzt Riquet. Riquet. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να συγχαρώ την Κομισιόν για την ποιότητα τη παρουσίασή τη. Με ενδιαφέρει το θέμα γιατί εγώ ήμουν εισηγητή δύο φορές για την ασφάλεια σκάφη. Έχω δύο ερωτήσεις σε δύο επίπεδα. Εισήγατε ουσιαστικέ μεταρρυθμίσεις για την ε, σταθερότητα των σκαφών και το είπατε και στην παρουσίασή σα, για τα ROPAX, δηλαδή ένα πολύ σημαντικό τμήμα της συνολικής μετακίνησης και των σκαφών στην Ευρωπαϊκή Να γίνει καλύτερη διαμερισματοποίηση, να γίνουν μεγαλύτερα τα σκάφη, που σημαίνει όχι μόνο ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν με βαριά έργα τα σκάφη, αλλά θα πρέπει να μειωθεί ουσιαστικά η ταχύτητά τους σε ανταπόκριση προς ε, λιμενικές ε, διατάξεις ασφαλείας. Τώρα είπατε ότι συζητήσατε με τις αρχές, αλλά δεν καταφέρατε να συζητήσετε με τις ενώσεις επιβατών. Αλλά προφανώς δεν μιλήσατε και με τον κλάδο, ο οποίος ανησυχεί έντονα για τον ισχυρό αντίκτυπο, οικονομικό και άλλο, επί της προσαρμογής των ρόμπαξ. Επομένως, η ερώτηση καθότι έχετε ήδη υποβάλει την πρόταση στο Συμβούλιο και θα την προτείνετε και στον IMO φαντάζεστε προβλέπετε να το συζητήσετε με τον κλάδο σχετικά με τόσο σημαντικές μεταρρυθμίσεις διατάξεων που θα έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον κλάδο αυτόν που είναι σημαντικός για την Ευρωπαϊκή δηλαδή εγώ εκπλήσωμαι για τα ισχυρότατα αυτά μέτρα που προτείνονται χωρίς να έχουμε συζητήσει τον κλάδο. Προφανώς και συμφωνώ με τους συναδέλφους και επιθυμώ και εγώ μέτρα, αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τους επιβάτες. Θυμίζω βεβαίως ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη σταθερότητα των σε τα μέτρα ασφαλείας. Αυτά που δηλαδή μας αναφέρατε στην παρουσίασή σας. Πάντως ανησυχώ για την πρώτη τέτοιων μέτρων χωρί να έχει γίνει επαναλαμβάνω διαβούλευση με τον κλάδο. Παρά μόνο εκ των υστέρων. Καλύτερα να μιλούμε εκ των προτέρων. Επίσης, μάλλον επαναλαμβάνω την ερώτηση. Θα μιλήσετε με τον κλάδο κάποια στιγμή. Danke sehr, jetzt Bruno Gollnisch. Ευχαριστούμε. Μπρούνο Γκρόνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την ίδια ερώτηση ήθελα να υποβάλω όπως και ο κύριος ε, Αγκέ για τη διαβούλευση. Αυτός το έκανε πολύ καλύτερα από μένα. Δεν θα επανέλθω. Ήθελα επίσης να προσθέσω το δικό μου ερωτηματικό σχετικά με την μη εφαρμοσιμότητα από ό,τι φαίνεται της Ιερακής Νομοθεσίας στο Κόσα Κονκόρδια. Γιατί σε σχέση με διατάξεις που έχουμε για την σημαία εφόσον μεταφέρουμε επιβάτες εντός των υδα... υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη στιγμή κατά την οποία ο πλειοκτήτης είναι Ευρωπαίος θα έπρεπε να υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ενδεχομένως δεν κατενόησα καλά ότι τα κάτω των 24 μέτρων δεν εμπίπτουν σε ευρωπαϊκή νομοθεσία, αν κατάλαβα καλά. Όμω δεν κατάλαβα ποιες είναι οι προθέσεις σα εκεί. Να τα εντάξετε στην ενισχυμένη ή τροποποιημένη νομοθεσία ή να αφήσετε τα πράγματα ως έχουν. Τουρικότητα δηλαδή. Απορία. Ευχαριστώ. Danke sehr. Und jetzt, Frau Berg, haben Sie... Σας ευχαριστώ και τώρα, κύριε Μπέρκ, να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με την πρώτη. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αυτά τα πορίσματα που συγκέντρωσε. Στην έκθεσή μας έχουμε ένα κατάλογο ε, με τις δράσεις μας 2014-308 είναι το έγγραφο. Τι προτείνουμε καταρχήν για την απλοποίηση. Σε μια πρώτη φάση έχουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα υποβληθούν την επόμενη άνοιξη και θα υπαχθούν στην κανονική νομοθετική διαδικασία. Θα προτείνουμε να καταργήσουμε κάποιες επικαλύψεις ε, στα καθεστώτα ελέγχου και επιθωρήσεων. Θα διευκρινίσουμε στην υπάρχουσα οδηγία κάποιους ορισμούς, για παράδειγμα τα πλοία το κατά πόσο τα πλοία που είναι από αλουμίνιο θα εμπίπτουν στην κοινωτική νομοθεσία ή όχι. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποιους ορισμούς ε, για τις προϋποθέσεις καταγραφής των επιβατών, ε, όπως προβλέπει η ισχύουσα οδηγία που είναι όμως του 1998. Επίσης θα προτείνουμε να αποκλείσουμε τα επιβατικά πλοία που είναι κάτω των 24 μέτρων και που έχουν χαλίδινη κατασκευή. Θα προτείνουμε τον αποκλεισμό τους από την υπάρχουσα οδηγία, γιατί είναι μόνο 70 τα πλοία, δηλαδή λιγότερο από 1% των επιβατηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι μελέτες μας έχουν δείξει ότι είναι υπερβολικά επαχθείς οι προϋποθέσεις για τα πλοία αυτά. Ούτε βρίσκονται σε ίδιο επίπεδο ανταγωνισμού με τα μικρότερα επιβατηγά που πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κατασκευασμένα από άλλα υλικά πλην του χάλιβος. Αυτό προτείνουμε αποκλεισμό τους. Και επίσης θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το, τα υπάρχοντα συστήματα ηλεκτρονικής καταγραφής που ήδη είναι διαλειτουργικά και έχουν κατασκευαστεί σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια τη Θάλασσα, προκειμένου να είναι διαθέσιμε οι πληροφορίε αρμόδιε αρχέ σε περίπτωση ατυχήματο. Δηλαδή, δεν αλλάζουμε τι υποχρεώσει, απλώ λέμε στου ε, διάφορου φορεί ότι θα πρέπει να αποστέλουν τους πλήρεις καταλόγους ε, επιβατών ε, με τους αριθμούς των επιβατών το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να είναι πολύ εύκολα προσιτές οι πληροφορίες σε όλους. Επίσης, προτείνουμε την αναβάθμιση των, εθνικών, των διεθνών προδιαγραφών για την ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων και για το θέμα αυτό έχουμε ήδη στείλει σχετική πρόταση στο Συμβούλιο. Θα απαντήσω αργότερα επί της ουσίας στους κυρίους Ρικέ και Γκόλνης. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τη διαπαφή μεταξύ των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία ισχύει μόνο για τα επιβατικά πλοία που πραγματοποιούν εσωτερικά δρομολόγια, δηλαδή δρομολόγια μεταξύ ε, δύο ε, κρατών μελών ή στο εσωτερικό των κρατών μελών. Για τα μεγαλύτερα επιβατικά, γιατί έχουμε τρεις διαφορετικές ε, κατηγορίες, τέσσερις μάλλον, ABCD, ανάλογα με το μέγεθος, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ισχύει για τα σκάφη της πρώτης κατηγορίας, για τα πλοία της πρώτης κατηγορίας. Πρόκειται για νομοθεσία που συμπίπτει με τους κανόνες και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Οπότε, αν δείτε την περίπτωση του Κώστα Κονκόρντια που έπλεμε Ιταλική σημαία, ναι, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και το Κώστα Κονκόρντια ήταν ε, πλοίο κατηγορία Α, θα έπρεπε να εφαρμόζεται και στο Κώστα Κονκόρντια. Επί της ουσίας όμως, όλες οι προδιαγραφές έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Γιατί σχεδόν κανένα από τα μεγάλα επιβατικά πλοία και κυρίως τα κρουαζιερόπλια δεν φέρουν σημαίες ευρωπαϊκού κράτους μέλους. Ήταν σύμπτωση ότι το Κώστα Κοκόρντι έφερε ιταλική σημαία. Συνήθως τα κρουαζιερόπλια έχουν σημαία Μπαχάμας ή ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και επειδή ακριβώς ε, αυτές ε, οι επιχειρήσεις ε, είναι παγκόσμιες εμβέλειες και δεν είναι σε τα πορθμία οχηματαγωγά ε, επιβατηγά που πηγαίνουμε μεταξύ, κυκλοφορούν μεταξύ δύο χωρών μελών. Ακριβώς επειδή λοιπόν είναι διεθνή τα δρομολόγια των κροσγεροπλοίων, ο κατάλληλο φορέας είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακό Οργανισμός και σχετική νομοθεσία. Γι' αυτό έχει νόημα τέτοιε κατηγορίε πλοίων να εμπίπτουν σε διεθνεί προδιαγραφέ. Μην ξεχνάτε ότι ένας πλειοκτήτης μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει τη σημαία καταγραφής του πλοίου του. Αν εμείς λοιπόν ως Ευρωπαίοι θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό και να εφαρμόσουμε πιο δρακόντια καθεστώτα για όλες τις κατηγορίες των επιβατικών πλοίων, το πιο πιθανό που θα γίνει είναι οι πλειοκτήτες να αλλάξουν τις σημαίες των πλοίων τους και να μην φέρουν πια ευρωπαϊκές σημαίες για να αποφύγουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό δεν είναι δυνατό για τα μικρότερα πλοία και γι' αυτό ακριβώς έχουμε την οδηγία για τα ROPAX, για αυτά τα ferry boat απορθμία γιατί ε, δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δρομολόγια τους γίνονται μεταξύ ευρωπαϊκών λιμένων. Για τα υπεροκειάνια όμως και τα κουρασγερόπλια έχει νόημα η ρύθμιση να είναι διεθνής, να εμπίπτουν σε διεθνή νομοθεσία. Τώρα, τι θα υπαχθεί σε διεθνή νομοθεσία. Το, αυτός ε, για τη δευτάθεια και την ασφάλεια του πλοίου σχετίζεται με τη διαμερισματοποίηση του πλοίου, όπως είπε ο κύριος Ρικέ. Και μετά το, το ναυάγιο του Εστόνια έχουν θεσπιστεί κανόνες σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που προβλέπουν ότι ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών και το μέγεθος του πλοίου θα απαιτούνται τόσο διαμερίσματα, τόσο διαφορετικά. Οπότε όταν το σκάφος υποστεί βλάβη να μην πλημμυρίσει ολόκληρο το πλοίο. Και αυτός είναι ένας τρόπος ε, θέσπιση νομοθεσία, αλλά υπερβολικά κατηγορηματικό και δεν ενισχύει και την καινοτομία. Γι' αυτό και το 2009 ο IMO τροποποίησε του διεθνεί κανόνε και είπε ότι εμεί τώρα προβλέπουμε διαφορετική προσέγγιση που θα είναι πιο φιλική προ την καινοτομία και θα αφήνει στο σχεδιαστή να αποφασίσει πόσα στεγανά θα έχει μέσα στο πλοίο, πόσα στεγανοποιημένα διαμερίσματα, ώστε να μπορεί το πλοίο να πλέει ε, και μετά την καταστροφή τμήματος του σκάφους του. Και οι νέοι κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού προβλέπουν ότι ένα πλοίο θα πρέπει να επιπλέει ε, και μετά από πολλά σενάρια καταστροφής, αλλά να πόκειται στο σχεδιαστή του πλοίου ε, να αποφασίσει ότι θα επιπλέει ακόμη και μετά από 80%, 95% ζημίας του σκάφους, για να μην υπάρχει το, ο κίνδυνος της ανατροπής ε, ή του ναυαγιού, ακόμη και μετά από σημαντική βλάβη του σκάφους. Οπότε αυτό συνέβησαν το 2009. Οπότε έκτοτε, ε, επειδή και εμείς θεωρούμε ότι η προσέγγιση αυτή είναι καλή και συνάδει με την καινοτομία, γιατί θέλουμε να μην είμαστε ε, πολύ κατηγορηματική και αποκλειστική και να αφήνουμε και χώρο και στην καινοτομία. Και έτσι μετά το 2009 όταν ε, εφαρμόστηκε αυτή η διεθνή νομοθεσία και αφορά το καθεστώς για τη σταθερότητα και την εφτάση μάλλον των ferry boats σε περίπτωση κατασκευής και ακριβώς επειδή τέτοια απορθμία κινούνται μεταξύ ευρωπαϊκών ε, λιμανιών ε, φροντίσαμε να ελέγξουμε κατά πόσο οι νέοι κανόνε του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού είναι εξίσου καλοί με του παλιού. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε εκπόνηση μελετών. Και τα τελευταία 15 χρόνια ε, και μάλιστα και μετά το 2009 έχουμε δαπανίσει περίπου τα 4 εκατομμύρια ευρώ στις μελέτες που έχουμε δώσει ε, στους, στον κλάδο, στους εφοπλιστές, στους σχεδιαστές για να μελετήσουν κατά πόσο με βάση τους νέους κανόνες μπορούν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν πλοία που θα είναι πιο ασφαλή. Δηλαδή δεν θα βουλιάζουν τόσο γρήγορα σε περίπτωση που το σκάφος τους έχει καταστραφεί, έχει υποστεί ζημίες. Βέβαια μετά από τις μελέτες καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πολλά μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί η δυνατότητα ε, επιβίωσης ε, ενός πλοίου, μην ε, ανατροπής δηλαδή σε περίπτωση που καταστραφεί ένα τμήμα του σκάφους. Και βέβαια δεν θέλησαμε να αναγκάσουμε τον τομέα να αλλάξει το επιχειρησιακό μοντέλο και σε ό,τι αφορά την ερώτηση κατά πόσο είχαμε διαβουλεύσει με τον κλάδο, ναι, είχαμε. Νομίζω ότι έτσι κάλυψα τα ουσιώδη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και πάλι για την παρουσίαση. Ήταν εξαιρετική παρουσίαση, αλλά από τα 45 λεπτά τα οποία είχαμε στη διάθεσή μα, ε, ξοδεύσατε τα 35. Ε, ήταν μικρή η συνεισφορά του Κοινοβουλίου, γιατί ουσιαστικά εμεί θέλαμε να γίνει συζήτηση. Την άλλη φορά σας παρακαλώ λοιπόν να, να τηρήσετε τα χρονικά όρια για να έχουμε επαρκή χρόνο και για τη συζήτηση μετά. Και περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Das ist der Bericht zum Absturz. Μιλάμε για την έκθεση σχετικά με τη συντριβή του MH17, συζήτηση με τον κύριο Έρβιν Μιούλερ, αντιπρόεδρο του Ολλανδικού Συμβουλίου Ασφαλείας, τον κύριο Πατρική. Να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα στο Σπνάι. Δεν ήταν λάθος του πιλότου και δεν έχει ακόμα διαλευκανθεί. Αλλά ακόμα και η προκαταρτική αυτή διαλευκανσή καταδεικνύει τη δυσκολία και την περιπλοκότητα της κατάστασης. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα... Καθίστε παρακαλώ. Und begrüße recht herzlich Herrn. Dutch Safety Board, και τον κύριο Πατρική, εκτελεστικό διευθυντή της ΑΕΔ. Und wie Sie wissen, hat der Dutch Safety Board am 13. Και όπως ξέρετε, χτες στις 13 ε, Οκτωβρίου παρουσίασε και δημοσίευσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, τα πορίσματά του για την ε, δυστύχημα του MH17. Έχασαν τη ζωή τους 298 επιβαίνοντες, οι πιο πολλοί από τους οποίους ήταν Ολλανδοί, Ολλανδικής υπηκότητας και παρά το γεγονό ότι το δυστύχημα έγινε στον αέριο χώρο της Ουκρανίας, η Ουκρανία, η κυβέρνηση της ε, Ουκρανίας έδωσε την αρμοδιότητα έρευνας ε, του δυστυχήματος στις κάτω χώρες της Ολλανδίας και συμμετείχαν και εκπρόσωποι από την Μαλαισία και από άλλες χώρες, καθώς και εμπειρογνώμονες από την Ουκρανία, τη Μαλαισία, της ΗΠΑ, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία. Και από τα στοιχεία προκύπτουν οι καταστάσεις και έτσι α, διαπιστώνουμε τι έγινε στην τραγωδία. Αυτή την τραγωδία την οποία συζητήσαμε συχνά ε, στην ε, Επιτροπή μας. Και γι' αυτό ζήτησα λοιπόν και από τον κύριο Πατρική, ε, εκλεστικό διευθυντή της ΕΕΔ, να παραστεί εδώ και να μας πει τι καινούριο υπάρχει σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας στην αεροπορία. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μιουλερ και μετά και στον ε, κύριο Κι για μια σύντομη προσθήκη. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση να μιλήσω εδώ και να σας εξηγήσω τα απορρίσματα της ε, ε, έρευνας και θα συνεχίσω τώρα στα Ολλανδικά. Κυρίε ε, και κύριοι. Ναι, ναι, ναι. Να το κάνετε, γιατί έχουμε και τερμηνία, λέει ο πρόεδρος, το ξέρω, το ξέρω. Κυρίε και κύριοι, στι 17 Ιουλίου 2014 η πτήση MH17 συνετρίβει στο ανατολικό τμήμα τη Ουκρανία. Η συντριβή και ο θάνατο 298 επιβαίνοντων ε, σώκαρε όλο τον κόσμο και έπληξε εκατοντάδε οικογένειε. Ε, τώρα, πριν από τέσσερι εβδομάδε, την 3η 13 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας της ε, Ολλανδίας δημοσίευσε την τελική εκθέση με τα πορίσματα σε σχέση με την έρευνα για τη συντριβή της πτήσης MS-17. Αυτό ασφαλώς και το ε, λάβατε υπόψη. Και σήμερα λοιπόν βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας για να παρουσιάσω τα απορρίσματα και να απαντήσω ενδεχόμενες ερωτήσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτελεί ανεξάρτητη αρχή ερευνητική της στην Ολλανδία που ερευνά τέτοια συγχήματα για να εξαγάγει τα συμπεράσματα προς την ασφάλεια και το μέλλον. Τους τελευταίους μήνες μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου ε, συμμετείχα ε, ε, πολύ στενά στις έρευνες για την συντριβή της πτήσης. Σε τέσσερα σημεία επικεντρωνόμαστε πώς εκτελήχθηκαν τα περιστατικά, η δρομή πτήσης, ο αντίκτυπος τους επιβαίνοντες και η δημοσίευση των στοιχείων των επιβατών. Και στην παρουσίαση αυτή θα επικεντρωθώ στα πώς εκτελέχθηκαν τα περιστατικά και στη διαδρομή της πτήσης, της πτήσης MH17 ε, πάνω από μία περιοχή σύγκρουση, γιατί πιστεύω ότι αυτά αφορούν το Κοινοβούλιο και επειδή οι εικόνε μιλούν πιο πολύ από χίλιε λέξει, θα ήθελα να σα δείξω και δύο μικρά βίντεο. Καταρχά, θα κοιτάξουμε τη συντριβή και την τάιτα της συντριβή στι 17 Ιουλίου 2014 στι 15 και 20 ώρα Ολλανδία στερματίστηκε απότομα η πτήση MH17 και οι 298 επιμένοντες έχασαν τη ζωή τους. Και το Συμβούλιο Ασφαλείας έκανε ειδικέ ερεύνες, έκανε και μια αναπαράσταση της συντριβής για να βρει τις αιτίες της συντριβής. Τρεις είναι βασικές αιτίες. Η πτήση MH17 συντριβή για την εξωτερική πλευρά πάνω από το αριστερό τμήμα του cockpit ε, εξεράγει ένα βλήμα. Αυτή η κεφαλή λοιπόν είναι τύπου του 9N314M και ε, τοποθετείται πάνω σε πύραυλο σε βλήμα όπως ε, σε βλήμα εδάφους αέρος BOOK. Είναι νομίζω πολύ κρίσιμο αυτό ως πόρισμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν της έκρησης είναι ότι έσπασε το πρόσθετο τμήμα του αεροσκάφους και έτσι διαλύθηκε στον αέρα το αεροσκάφος. Ε, και τα συντρίμια έπεσαν σε μια περιοχή 50 ε, ε, τετραγωνικών χιλιόμετρων στην ανατολική πλευρά της Ουκρανίας. Το βλήμα λοιπόν επίσης ε, προήλθε από μια ε, περιοχή 300 320 τετραγωνικών χιλιόμετρων στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Και ας δούμε λοιπόν το πρώτο βίντεο. We need some. Geluid. Start again maybe.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 Eh, eh, eh, Κυρίε και κύριοι, δεν έχουμε τον ήχο και άρα θα σας δώσω εγώ κάποια σχόλια. Βλέπετε λοιπόν την DCMH 17 στι 17 Ιουλίου 2014, προορισμός Παλαλουμπούρ. Ε, περνάει τα από την περιοχή. Έχει υπάρχει ε, νέφωση περνάει πάνω από την Ουκρανία λοιπόν, όπου ε, μεγάλο τμήμα του ενέργου χώρου είναι κλειστός, μέχρι τα 20.000 πόδια και πάνω από τα 300.000 πόδια ε, είναι η διαδρομή την οποία διανύει το MH17. Μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο αυτά ως αναπαράσταση. Τη στιγμή λοιπόν στις 15 και η 20 εκτοξεύεται πύραυλος από ένα σύστημα εκτόξευσης BOOK, εδάφους αέρους, οποία, το οποίο βλήμα και ε, εκρήγνεται κοντά στο αεροσκάφο. Και ε, το βλήμα λοιπόν αυτό περιλαμβάνει διάφορα υποστοιχεία, τα βλέπετε. Υπάρχει, ε, υπάρχουν αυτά τα α, στοιχεία τα οποία προσωμιάζουν σε σχήμα πέτα τα οποία και βρήκαμε μέσα στο κόκπιτ και στους πιλότους. Βλέπετε λοιπόν πόσο το βλήμα πλησιάζει το αεροσκάφος και πώς χτυπάει αριστερά στο κόκπιτ και στη συνέχεια λοιπόν συνετρίβεται, διερυκνύεται το αεροσκάφος, πέφτει το κόκπιτ και έτσι συνετρίβει όλο το αεροσκάφος στον αέρα. Και τα συντρίμια λοιπόν πέφτουν το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Αυτά ήταν τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν στην αναπαράσταση αυτή και βλέπετε λοιπόν κάποια από τα συντρίμια τα οποία κατέληξαν στο έδαφος. Βλέπετε λοιπόν και τα συμπεράσματα τα οποία μόλις σας ανέφερα. Στα 33.000 πόδια πετούσε το αεροπλάνο η πτήση ε, εκτήλησε όταν κανονικά δεν υπήρχαν προβλήματα ούτε με το πείραμα ούτε με τους πιλότους, δεν υπήρχε κανένα μήνυμα ε, από το cockpit. Βρήκαμε και το voice recorder του cockpit αλλά και άλλο recorder οπότε και μπορέσαμε να αναλύσουμε σωστά τα στοιχεία και στις 13 ε, και σταμάτησαν οι καταγραφές. Ε, υπήρξε λοιπόν ε, διάτρηση από πολλά και ξεχωριστά σωματίδια. Κάναμε λοιπόν μια αναπαράσταση ακριβή στις κατοχώρες και βλέπετε λοιπόν ποια ήταν τα σωματίδια αυτά, πώς έγινε και η αναπαράσταση αυτή, η οποία και ξεκαθαρίζει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι αυτή ήταν η αίτια του δυστυχήματος και βλέπετε λοιπόν τώρα και στο βίντεο ότι βρήκαμε και κάποια τμήματα πυράβλου που ταιριάζουν με αυτά που βρέθηκαν στο αεροσκάφος. Κάναμε και μία ανάλυση των όσων ακούσαμε από το κόκπιτ, από τα διάφορα μικρόφωνα και αυτό ε, ταιριάζει με μία εξωτερική ε, έκρηξη. Και βλέπετε λοιπόν πως ε, έσπασε το αεροσκάφο σε έξι διαφορετικά κομμάτια και βρέθηκαν λοιπόν τα συντρέμια αυτά στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Εκτόξευση λοιπόν του πυράβλου, έκρηξη στο, άνατο, στο αριστερό τμήμα του κόκπιτ τα τρία άτομα μέσα στο κόκπιτ ε, έχασαν τη ζωή τους ε, πάρα αυτά. Οι υπόλοιποι επιβάτε έχασαν τη ζωή του μετά από ένα, ένα μισή λεπτά. Όλοι οι επιβαίνοντε έχασαν τη ζωή του λοιπόν, όταν το αεροπλάνο συνετρίβει στο έδαφο. Αυτά, λοιπόν, ήταν τα σχόλια από δική μου πλευρά. Αμέσω μετά το δυστύχημα λοιπόν της πτήσης MH17 ήταν σαφέ ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έπρεπε να συμβάλλει στην έρευνα του τι συνέβη και την ίδια ημέρα μετά το δυστύχημα οι ερευνητέ μας πήγαν στην Ουκρανία για να συνδράμουν. Στις 23 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο Ασφαλεία ανέλαβε την ηγεσία της διεθνούς έρευνα για τα περιστατικά της δυστυχήματος. Και αυτό έγινε μετά από αίτηση των Ουκρανικών αρχών, γιατί για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε τα ακριβή περιστατικά της συντριβής όπως γίνεται σε μεγάλα αεροπορικά δυστυχήματα. Αυτό τι σημαίνει, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές της έρευνας για τέτοια δυστυχήματα που ορίζονται στο παράδειγμα 13 της Σύμβασης του Σικάγο. Επτά χώρες λοιπόν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, συμμετείχαν ως ε, διαπιστευμένοι εκπρόσωποι στην έρευνα αυτή. Η Ολλανδία, η Ουκρανία, η Μαλαισία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, η Ηνωμένο Βασίλεια, η Αυστραλία και η Ρωσική Ομοσπονδία. Και στο πλαίσιο του ΙΚΑΟ ε, φάνηκε ότι αυτή η έρευνα είχε μεγάλη αξία. Αποτέλεσε τη βάση μια καλή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών και κατέστησε δυνατή την διεξαγωγή, την εξαγωγή πορισμάτων με του εκπρόσωπους των χωρών που ε, συμμετείχαν. Και αυτό ασφαλώς ε, καθόρισε και την ποιότητα της έρευνας. Η δεύτερη λοιπόν έρευνα επικεντρώθηκε στη διαδρομή πτήση. Κυρίω γιατί πετούσε η πτήση των Malaysia Airlines των Μαλαισιανών αερογραμμών MH17 πάνω από μια περιοχή σύγκρουση, ε, όπου εκείνη την ε, στιγμή υπήρχε ένοπλη σύραξη. Είναι μια ερώτηση που απασχόλησε πάρα πολλού και απασχολεί ακόμα πάρα πολλού. Ε, η απάντηση είναι αρκετά απλή αλλά και πολύ Μα προκαλεί μεγάλο προβληματισμό γιατί όλοι ουσιαστικά πετούσαν πάνω από την περιοχή και γιατί, γιατί κανείς δεν θεωρούσε ότι διατρέχαν κίνδυνο οι πολιτικέ πτήσει. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν ποιε περιο... και διερευνήσαμε αμέσω ποιε αεροπορικέ εταιρείε πετούσαν πάνω από την περιοχή αυτή μεταξύ 14 και 17 Ιουλίου 2016. Μία αεροπορικές εταιρείε, 61 εταιρείε από 32 διαφορετικές χώρες και την ημέρα λοιπόν του δυστυχήματο. 160 πτήσεις πέρασαν από το ανατολικό τμήμα αυτό της Ουκρανίας μέχρι να κλείσει ο εναωρίας χώρος αυτός. Όλοι σχεδόν λοιπόν πετούσαν εκεί σχεδόν. Και όλες οι αεροπορικές εταιρείες θεωρούσαν ότι ήταν και ασφαλείς οι πτήσεις αυτές. Ε, γιατί μπορεί να υπήρχε ε, στο έδαφος η σύγκρουση, αλλά ο εναέριος χώρος πάνω από τα 32.000 ε, πόδια, 10 περίπου χιλιόμετρα, δεν ήταν ανοιχτός για τις πολιτικές πτήσεις. Κανείς δεν θεώρησε ότι οι πτήσεις, οι πολιτικές πτήσεις σε ύψος πλεύσης θα μπορούσαν να διατρέχουν κίνδυνο. Στη σύμβαση του Σικάγο, τη Διεθνή Σύμβαση για θέματα πολιτικών ε, πτήσεων, αναφέρεται ότι είναι ευθύνη του κράτους να καθορίσει κατά πόσον ε, ενήρος χώρος πάνω από την επικράτειά του είναι ασφαλής ή όχι. Τις ε, μήνες λοιπόν πριν από το δυστύχημα, 16 ήταν τα στρατιωτικά αεροπλάνα και ελικόπτερα που καταρρίφθησαν τον ανατολικό τμήμα τη Ουκρανία. Και αυτό το ήξεραν οι ουκρανικέ αρχέ και δήλωσαν ότι σε κάποιε περιπτώσει χρησιμοποιήθηκαν και οπλικά συστήματα τα οποία μπορούσαν να φτάσουν σε ύψο πλεύση. Παρ' όλα αυτά όμω η Ουκρανία δεν είχε κλείσει τον αέριο χώρο τη. και η Ουκρανία ε, διατείνεται ότι δεν υπήρχαν επαρκεί ε, ενδείξει για να κλείσουν τον αέριο χώρο στην ανατολικά τη χώρα. Ε, το δικό μα πόρισμα είναι διαφορετικό. Το δικό μα πόρισμα είναι ότι υπήρχαν επαρκεί ενδείξει για να κλείσουν προοπτικά οι Ουκρανικέ αρχέ στον αέριο χώρο του σε ό,τι αφορά το ανατολικό τμήμα αυτό τη χώρα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η Ουκρανία ω κράτο, αλλά και όλε οι αεροπορικέ εταιρείε και άλλε χώρε και οι μυστικέ υπηρεσίε και οι διεθνεί οργανώσει οι διεθνεί οργανισμοί δεν αξιολόγησαν με σωστό τρόπο τον κίνδυνο για του πολίτε. Και από την έρευνά μα προκύπτει ότι όλα τα, όλοι οι φορείς με φυσική διάσταση κοιτούσαν πολύ προσεκτικά την, ε, ε, τα ανατολικά τη Ουκρανία. Αλλά κανείς δεν θεωρούσε ότι ήταν κίνδυνο για τι πτήσεις, τις πολιτικές πτήσεις. Έχουμε λοιπόν κάποια σαφή διδάγματα να αντλήσουμε και τα πορίσματά μας έχουν να κάνουν ουσιαστικά αποκλειστικά με τις διαδρομές πτήσης. Χρειάζονται λοιπόν μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων και θα ήθελα να κάνω τριών ειδών συστάσεις. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι είναι σημαντικό να είναι πιο δεσμευτική και πολύ πιο αυστηρή η διαμόρφωση της ευθύνη του κυριαρχού κράτου για τον αέριο χώρο του. Θα πρέπει να είναι σαφές το πότε και υπό ποιου όρου θα πρέπει να κλείνει ένα κράτος στον αέριο χώρο του και θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση στο πώς τα κράτη και οι αεροπορικές εταιρείες εκτιμούν τους κινδύνους σε ό,τι αφορά πτήσει πάνω από περιοχές συγκρούσεων. Όσο πιο γρήγορα γίνεται θα πρέπει να δίδονται πληροφορίε για τέτοιε ένοπλε συγκρούσει και αυτέ θα πρέπει να ανατίθενται σε όλου που είναι υπεύθυνοι για λήψη τέτοιων αποφάσεων για τι δρομέ πτήση. Και τέλο, πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αεροπορικέ εταιρείε να είναι διαφανεί και προ το κοινό σε ό,τι αφορά τις πτήσεις, ε, τις διαδρομές πτήσεων που ακολουθούνται για να ξέρουμε κι εμεί ω πολίτε, ω επιβάτε ποια ε, διαδρομή θα ακολουθήσει κάθε για να μπορούμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα αυτά θα πρέπει να προσαρμοστεί και η διεθνή νομοθεσία για να αεροπορία το Συμβούλιο Ασφαλείας των Καταχωρών πιστεύει ότι θα πρέπει και τα κρατημέλη και οι μυστικές υπηρεσίες, οι αεροπορικές εταιρείε και οι διεθνείς οργανισμοί να διαμορφώσουν από κοινού τέτοια μέτρα για τις πτήσεις πάνω από περιοχές συγκρούσεων. Και ελπίζουμε ότι οι συστάσεις οι οποίες θα απευθύνουμε προς τα κράτη θα μπορέσουν να ακολουθηθούν από όλα τα κράτη. Τέλος, ε, πρόεδρε, και θα ολοκληρώσω στο σημείο αυτό. Η ε, έρευνά μας έλαβε χώρα υπό πολύ ιδιαίτερε συνθήκε. Δεν μπορούσαμε να πάμε και να ερευνήσουμε ε, απλά γιατί δεν μας έδωσαν και όλες τις πληροφορίες και φυσικά ε, μας πήρε και πάρα πολύ χρόνο να συγκεντρώσουμε όλα τα συντρέμια στις κάτω χώρες και αυτό δεν το αγνοήσαμε αλλά προσπαθήσαμε να προστασιοποιηθούμε στο βαθμό του δυνατού από τη διεθνή και εθνική πολιτική γιατί αυτό που ήταν βασικά για μας και για τα συμπεράσματά μας ήταν τα πραγματικά περιστατικά οι διάφορες αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές θεωρούμε ότι έχουν καθήκον να αντλήσουν διδάγματα από το δυστύχημα αυτό και να ηγηθούν της προσπάθειας για την τροποποίηση της νομοθεσίας και ελπίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή να δραστηριοποιηθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μούλερ. Και τώρα το λόγο έχει ο κ. Κι για να κάνει τις προσθήκε. Vielleicht noch bevor wir anfangen möchte ich. ξεκινήσουμε, λέει ο Πρόεδρο, θα ήθελα να καλωσορίσω μία ομάδα επισκεπτών στην Επιτροπή μα. Ε, πέντε λοιπόν επισκέπτε ε, τη κυρία Γκράσμαν ε, από την Βιέννη. Und jetzt, Herr Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. my Εγώ δεν θα σχολιάσω τα πορίσματα της έρευνας που παρουσίασε ο Ολλανδός συνάδελφος αλλά θα αναφερθώ στις διάφορες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αναλάβαμε μετά από την τραγωδία αυτή. Καταρχά να δούμε, να έχουμε μία εικόνα των απειλών. Παρουσιάστηκαν πλήρως από τον Ολλανδό συνάδελφο. Με το δυστύχημα αυτό αναδείχθηκε μία νέα τάξη απειλής με αυτά τα με αυτούς τους πυράβλους εδάφους αέρας για την κατάρριψη αεροσκαφών επιβατηγών που είναι αντιπροσωπεύει μια νέα απειλή αλλά έχουμε και άλλες αντίστοιχες φύσεως όμως διαφορετικές ως προς τις μεθόδους έχουμε αυτό που ονομάζουμε manpad ένα μικρή εμβέλειας εδάφους αέρος πυροβόλο ατομικό και είχαμε και κάποια ατυχήματα με τέτοια στο παρελθόν. Και έχουμε και άλλου είδους απειλές, όπως είχαμε δει και φέτος τον Οκτώβριο, με πυράβλους cruise που είχαν εκτοξευθεί από την ε, Κασπία 27 πύραυλοι διέσχισαν ενέριο χώρο χώρο στον οποίο κινούνται επιβατικά αεροσκάφη. Και ενημερωθήκαμε για την εκτόξευση των πυράβλων αυτών από αναφορές σκαφών που πετούσαν στην περιοχή αυτή and πειρατικών σκαφών λέει ο μιλητής που πετούσαν στην περιοχή και τον Οκτώβριο επίσης η Ρωσική Ομοσπονδία ζήτησε απολύτως νόμιμα υπό τις διεθνείς συμβάσεις να κλείσει ενέργειος χώρος στη, Μεσογειακή Λεκάνη νοτιοανατολικά της ε, Κύπρου προκειμένου να πραγματοποιήσουν δοκιμές ε, εκτόξευσης πυράβλων. Ε, αυτή η περιοχή δεν είναι μια περιοχή πολεμικής σύγκρουσης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δοκιμή, για τη δοκιμαστική χρήση πυράβλων που είναι απειλή για την ε, αεροπλοεία. Λοιπόν, από το 70 είχαμε 33 δυστυχήματα με 1500 ε, θύματα αεροσκαφών. Κυρίως, κυρίως από manpads, από ατομικά τέτοια πυροβόλα όπου εκτοξεύεται ένα βλήμα από τέτοιου είδους όπλο 18 είχαμε τέτοιες περιπτώσεις αλλά είχαμε και είτε εδάφους αέρος είτε αέρος αέρος πυράβλους και βλήματα που χρησιμοποιήθηκαν ή στην περιοχή των επιβατικών αεροσκαφών. Εν πάση περιπτώσει δεν μιλούμε για έναν μικρό αριθμό για τα τελευταία 50 έτη, αλλά υπάρχει και μία συνέπεια συνολική που είναι ο αντίκτυπος επί των μεγεθών επιβατών, των αριθμών επιβατών. Αν κοιτάξουμε τους αριθμούς επιβατών από την Ευρωπαϊκή προς το Ντουμπάι ή προς την Νοτιοανατολική Ασία πολλές από αυτές τις πτήσεις διασχίζουν ένα αέριο χώρο πάνω από πολεμικές συγκρούσεις και το γεγονός ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την συντομότερη οδό, να λάβουν τη συντομότερη οδό αυτές οι πτήσεις έχει αντίκτυπο και οικονομικό αλλά βεβαίως και επί της ασφάλειας των επιβάτων. Λοιπόν, η ανάλυση μας είναι ότι υπάρχει απειλή επιθέσεων ή και κατά λάθο κρουσμάτων, βλημάτων ή πυράβλων που να εκτοξεύονται. Είχαμε και μικρά πυροβολά όπλα όπως καλάσινικοφ να πυροβολούν προς αεροσκάφη και έχουμε διάφορες κατηγορίες απειλής σε ενδιάμεσα και υψηλότερα υψόμετρα. Τώρα έχουμε προχωρήσει σε κάποιες δράσεις τις οποίες θα αναφερθώ αργότερα που ο αντίκτυπός τους ήταν να κλείσει συγκεκριμένη ζώνη εναερίου χώρου κάτω από τον οποίο υπήρχαν πολεμικές συγκρούσεις. Αυτό δημιουργεί με τη σειρά του προβλήματα συμφόρησης και οικονομικές συνέπειες σε κάποιες από τις χώρες από τις οποίες δεν περνούμε πλέον λόγω του πλησίματος εναερίων χώρων. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και μάλιστα αμέσως μετά το δυστύχημα ήταν να προβλέψουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό συναγερμού ψήματος εκτάκτου ανάγκης που να παρέχει ασφάλεια σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής να έχουμε μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών κινδύνου που να διατίθεται για όλους τους ε, αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς, αρχές εταιρείε και επιβάτες. Και προχωρήσαμε σε μια αξιολόγηση κινδύνου για τις ε, επικίνδυνες ζώνες πολεμικών συγκρούσεων. Μια τέτοια αξιολόγηση κινδύνου αναφέρθηκε και ο προηγούμενο ομιλητή Εξαρτάται εν πολλή από την εντύπωση που έχει κανείς για το κίνδυνο. Για, το, για παράδειγμα, το 2014 είχαμε ένα σήμα για το αεροδρόμιο του Μπεν στο Ισραήλ. Για την κυβέρνηση του Ισραήλ ο κίνδυνος ήταν πολύ χαμηλός. Για εμάς, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για κάποιες άλλες χώρες, ο κίνδυνος αξιολογήθηκε ως υψηλός. Αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν είναι να έχουμε κάποιες κοινέ παραμέτρους αξιολόγησης κινδύνου ώστε να δίνουμε στους αερομεταφορείς ένα επίπεδο χαμηλό, μέσο ή υψηλό κινδύνου. Γιατί τελικώς αυτό που επιχειρούμε είναι να έχουμε κοινή πληροφόρηση και κοινέ συστάσεις ενδεχομένω. προς τους αερομεταφορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Και πρέπει να είμαστε σε θέση να ενεργοποιούμε αυτές τις επικοινωνίες ταχύτατα. Και για να αναφερθώ ξανά στην Κασπία, η εκτόξευση των πυράβλων έγινε εντός 6 ωρών και έπρεπε να αντιδράσουμε σε ζωντανό χρόνο, όπως λέμε. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε εβδομάδες προτού δώσουμε πληροφορίε στους αερομεταφορείς και μάλιστα μετά από αυτό είχαμε αρκετούς αερομεταφορείς που ζητούσαν από εμάς τι πληροφορίες υπήρχαν και τι επρόκειτο να κάνουμε. Άρα λοιπόν, από το δυστύχημα του MH17, της πτήσης, τι έγινε. Προχωρήσαμε σε μια ενεργό ανάλυση των κινδύνων ζώνων σύγκρουσης όπως και σήματα κινδύνου που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές για τους δικούς τους αερομεταφορείς το οποίο έγινε από τρεις χώρες Ηνωμένε Πολιτείε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Και πολύ πρόσφατα το έκανε και η Γερμανία αυτό. Η ΑΙΚΕΟ, ο Διεθνής Οργανισμός, προχώρησε στη δημιουργία ενός task force με την εντολή να δημιουργηθεί ένα αρχείο, ένα μητρό για όλες τις εναέριες ζώνες που κλείνουν σε όλο τον κόσμο για λόγους κινδύνου. Η Κομισιόν και κυρίως η ΓΔ ΜΟΥΒ με τα κράτη-μέλη και την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως προχώρησε σε μια συλλογή κοινών μεθοδολογιών προκειμένου να αξιολογείται σε ποιες περιοχές του κόσμου έχουμε υψηλό κίνδυνο και για να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή κατανόηση για το επίπεδο αυτού του κινδύνου. Σε ό,τι αφορά στην ΕΑΣΑ, εμείς προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων τους οποίους θα μπορούσαμε να καλούμε ταχαίως να ανταλλάσσουμε πληροφορίες επίσης ταχαίως και να προετοιμάσουμε τις αντιδράσεις ή τις προληπτικές μας ενέργειες σε σχέση με την αξιολόγηση του κινδύνου που έχουμε κάνει για κάθε περιοχή. Δημοσιεύσαμε επίσης κάποια, κάποιες εκθέσεις ενημέρωσης ασφαλείας όχι μόνο για τους αερομεταφορείς αλλά για τη διεθνή κοινότητα όταν εκδίδεται συγκεκριμένο σήμα από συγκεκριμένη χώρα. Και εδώ στην διαφάνεια αυτή έχετε ένα κατάλογο αυτών των ε, δελτίων ενημέρωσης ασφαλείας που έχουμε δημοσιεύσει τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ακόμα ενεργά και εδώ τα βλέπετε και στο χάρτη δεν είναι έκπληξη που βλέπουμε μια πυκνότητα κινδύνου προς την Μέση Ανατολή και την Αφρική αλλά βεβαίως και την Ουκρανία ιδίως δε την Ανατολική Ουκρανία Τώρα οι προκλήσεις όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής δεν υπάρχει συνολική πληροφορία, συνολική πληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κίνδυνο είναι κατακαιρματισμένη η πληροφορία αυτή, βρίσκεται σε διάφορα σημεία, σε διάφορους φορείς και δεν κοινοποιείται αναγκαστικά προς το σύνολο των ενδιαφερομένων. Έχουμε διάφορους φορείς, δεν έχουμε ενιαία αλυσίδα λήψης απόφασης, έχουμε ακόμα αρκετές χώρες που ακολουθούν μια πολύ εθνική προσέγγιση απέναντι σε τέτοια επεισόδια ακόμα και ως προς τις εντολές που δίνουν προς τους δικούς τους αερομεταφορείς. Και το πρόβλημα είναι ότι οι Ευρωπαίοι επιβάτες δεν πετούν αναγκαστικά, αναγκαστικά λέει ο μιλητής, με τον εθνικό τους αερομεταφορέα. Επομένως, ποιος είναι ο στόχος, να προστατεύσουμε τους αερομεταφορείς ή τους επιβάτες ποιο είναι το ενδιαφέρον που έχουμε για να μοιραζόμαστε αυτές τις εντολές. Και σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς υπάρχουν κέντρα πληροφοριών και ανάλυσης, αυτά κυρίως σε στρατηγικό επίπεδο, δηλαδή αρκετούς μήνες εκ των προτέρων, αλλά όλες αυτές οι προσπάθειες εξαρτώνται εν πολλής από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα δίκτυο πληροφοριών ή μια υπηρεσία πληροφοριών. Εξαρτάται από τις πληροφορίες των κρατών μαλλών και το κατά πόσο τα κράτη-μέλη θέλουν να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες. Και καθότι ε, έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ανταλλαγή πληροφοριών και στον συντονισμό των ε, δράσεων που απαιτούνται για να έχει κανείς μια συνολική εικόνα. Όπως και στο επίπεδο της συνεργασίας που χρειάζεται για να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση επί τη βάση πορίσματος πληροφορίας δηλαδή. Επίσης οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών ε, δεν έχουν ως εντολή να μοιράζονται τις πληροφορίες που έχουν διαθεσί τους με το ευρύ κοινό και καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει διστακτικότητα, για να την πούμε έτσι, και εθνικά και βεβαίως διεθνώς. Δύο ακόμα λόγια, αν μου επιτρέπετε πρόεδρε, στην ΕΑΣΑ έχουμε ένα μικρό αριθμό χωρών που αμφισβητεί την αρμοδιότητα, να την πούμε έτσι, της ΕΑΣΑ σε αυτή την περιοχή, γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Όμως αυτό το ζήτημα ε, τίθεται ρητορικά, γιατί στο τέλος τέλος είναι η ζωή των επιβατών που απειλείται και κάποιος πρέπει να αναλάβει δράση. Θα έλεγα λοιπόν συμπερισματικά το εξή. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, έχουμε συστήσει αυτήν την task force με εκπροσώπους των αερομεταφορέων, των εθνικών αρχών, των υπηρεσιών πληροφοριών και των ερωαϊκών θεσμών προκειμένου να βρούμε ένα τρόπο καλύτερης ανταλλαγής της πληροφορίας με τους κατάλληλους και αρμόδιους. Σα ευχαριστώ κύριε και τώρα ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσε και οι δύο παρουσιάσει που ακούσαμε και τώρα το λόγο έχει καταρχά ο Βιν Φαντεκάμπ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ πολύ μαζί σα ότι ότι και οι δύο παρουσιάσεις και οι δύο ιστορίες ε, που ακούσαμε σήμερα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές και συμφωνώ ότι το δυστύχημα την προηγούμενη εβδομάδα στην Αίγυπτο ανακοινεί και δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική στο δυστύχημα της πτήσης MH17. Έχω ένα αίσθημα κάθε φορά ότι εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και είμαστε ασφαλείς και κάνουμε τις συναντήσεις μας, αλλά ότι ο κόσμος ε, έξω είναι όλο και πιο απολυτικός και επικίνδυνος. Πέντε ερωτήσεις έχω να κάνω προς τον κύριο Μιούλερ και προς τον κύριο Κάι. Κι. Δεν ξέρω πώς προφέρετε το όνομά σας. Καταρχάς κύριε Μιούλερ, για τις, ε, τα, τις προειδοποιήσεις που υπήρχαν πριν, από πριν. Υπάρχει αστάθεια για τις ε, ενδείξεις, τις προειδοποιητικές, οι οποίες και αγνοήθηκαν, γιατί δεν λεφθήσαν υπόψη. Η άποψη της Eurocontrol ουσιαστικά είχαν προειδοποιήσει. Α, ναι, όχι. Ήταν δικό τους καθήκον να προβούν σε τέτοιες προειδοποίησεις. Δεύτερη ερώτηση για τα στοιχεία, τα δεδομένα των ραντάρ. Είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι το ήξεραν οι Ρώσοι ότι οι Ουκρανοί δεν είχαν ενεργοποιημένο ένα από τα συστήματα αυτά. Οι Ρώσοι μάλλον ε, είχαν διαγράψει τα στοιχεία αυτά και ο κύριος Κέρι από τη ΣΥΠΑ ανέφερε ότι απλά είδαμε ένα αεροσκάφος να πέφτει. Και επίσης, ποιος είναι ο ρόλος της ΙΚΑΟ, της Διεθνής, της Οργάνωσης ε, για την Πολιτική Αεροπορία. Ή έκανε κανείς ένσταση, προσφυγή προς τον ΙΚΑΟ για την απουσία των δεδομένων αυτών από ραντάρ. Τρίτη ερώτηση. Που συνδέεται και με την πρώτη υπήρχε ή δεν υπήρχε κατάλογος, λίστα αεροπορικών εταιριών που δεν πετούσαν πάνω από την Ανατολική Ουκρανία. Και εδώ επικρατεί μια μεγάλη ασάφεια. Κάποιες πετούσαν, κάποιες δεν πετούσαν. Και γιατί αυτές που δεν πετούσαν, δεν πετούσαν. Ε, δέστε τώρα δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Κι. Μας αναφέρεται το περιστατικό του Ισραήλ. πού είναι το καθήκον τη ΙΚΑΟ εδώ. Είπατε ότι χρειάζεται μια κοινή αξιολόγηση κινδύνου. Εγώ πάντα είχα την εντύπωση ότι αυτό το έκανε ήδη η ΙΚΑΟ. Γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τέλο Πρόεδρε, για τις μυστικές υπηρεσίε μία ερώτηση. Διαβάζοντας την ε, έκθεση για τις ρωσικές ε, υπηρεσίες και όσα γνωρίζουν οι Βρετανικές ε, μυστικές υπηρεσίες. Είναι όλα αυτά εντυπωσιακά. Αλλά βάση των μυστικών υπηρεσιών, όπως και στην αστυνομία, είναι το να κρατάμε τις ε, πληροφορίες ο καθένας για τον εαυτό του. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν. Άρα, το ερώτημα μου είναι το εξή. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασία τη ΕΑΖΑ με τι μυστικέ υπηρεσίε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτή η επικοινωνία από τις μυστικέ υπηρεσίε με τις άλλες οργανώσεις. Δηλαδή, ο κύριος Έρτοκ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μιούλερ και τον κύριο Κι για τις δύο αυτές παρουσιάσεις. Νομίζω ότι ο κύριος Κι μίλησε για το δίλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατεξοχήν. Είπατε ότι δεν υπάρχει ούτε μία αλυσίδα λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει δηλαδή να συμβεί προκειμένου τα κράτη-μέλη να σταματήσουν επιτέλου να κοιτάνε μόνο τα του οίκου τους. Δεν έχω αντιρρήσει ότι τα κρατη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν την καθημερινή τους ζωή αλλά τέτοια ζητήματα όπω η τρομοκρατία για παράδειγμα, τα οποία είναι διασυνοριακά, έμα δεν θα πρέπει να μεταφερθούν αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επανειλημμένα αναφέρθηκαν οι μυστικέ υπηρεσίε. Δεν θέλω να απαιτήσω τη δημιουργία μια Ευρωπαϊκή Μυστική Υπηρεσία, αλλά να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε. Και κοιτώντα τι, τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, ε, ο, ανησυχεί κανεί. κανείς ε, με τον αριθμό των στοιχημάτων. Στον νοτιοανατολικά της ε, Μεσογείου η Ρωσία θέλει να κάνει πειράματα με πυράβλους και λίγο πιο βόρεια ξέρουμε ότι υπάρχει η σύγκρουση μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας η οποία περιλαμβάνει όλο και πιο πολλά οπλικά συστήματα και ε, εδώ και μήνες στην Ευρώπη συζητάμε το θέμα της Ελλάδας, έχουμε γίνει παρανοϊκοί με τους πρόσφυγες. Ενώ γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξεσπάνε όλο και πιο πολλές κρίσεις. Θα πρέπει επιτέλους να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας των κρατών μελών. Μία ερώτηση προς την ΕΑΖΑ, προς την κύριο Κι. Αληθεύει, κύριε Κι. ότι πριν το δυστύχημα του MH17 υπήρχε μυστικές υπηρεσίες, βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, ένας πράκτορας ο οποίος ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να πετάνε αεροσκάφη πάνω από την περιοχή αυτή. Αν αληθεύει αυτό για την British Airways και αν οι μυστικέ υπηρεσίε τη Βρετανία το κράτησαν αυτό για τον εαυτό του, μπορεί να είναι νόμιμο αυτό, αλλά τελικά το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Αν αληθεύουν λοιπόν αυτά, καταδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία πέρα από τα εθνικά σύνορα. Η τρομοκρατία είναι κάτι καθολικό, παγκόσμιο, όπως και το κλίμα, για παράδειγμα, η προστασία του κλίματος. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τους πολίτες μας από τέτοια τραγικά περιστατικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει ο κύριος Κράμερ, η Τζάκη Φώστερ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους δύο καλεσμένους, τον εκπρόσωπο του ε, Ολλανδικού Διοικητικού Συμβουλίου Ασφάλειας και τον κυρίο Κι. Ε, Μάλιστα, εγώ εργάστηκα στον κλάδο αυτό και όταν ήταν συχνά φαινόμενο και αεροπειρατείες. Οπότε έχω γνώση του κλάδου και ευχαριστώ και τις Ολλανδικές Αρχές και όλους ε, εκείνους που συμμετείχαν ε, στην έρευνα που ήταν πολύ μεστή και μάλιστα υπό αντίξωες συνθήκες. Γιατί ε, μπορεί να μην ήταν τρομοκρατική επίθεση και μπορεί να μην ε, ήξερα αν ήταν μαλαισιανό πολιτικό αεροσκάφο Όπως και να έχει το πράγμα, πάντως ε, το κακό έγινε και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τώρα, κάτι πιο θετικό. Θα έλεγα ότι το θετικό σημείο για την πολιτική αεροπορία είναι ότι προσπαθούμε να φτάσουμε ε, στην ε, ουσία της κατάστασης, να δούμε τι πραγματικά έγινε και να αντιμετωπίσουμε και παγκοσμίω παρόμοια θέματα. Δεν θέλω να αναζητώ ενόχου. κανένα δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα καταρριφθεί το μαλαισιανό αεροσκάφο από πύραυλο. Και θα πρέπει να καταλάβουμε και το κοινό να το καταλάβει, ό,τι και να κάνουμε σε όποιο τομέα μεταφορών στηρίζεται στους κινδύνους. Και εγώ ε, πέταξα πολλές φορές από ζώνες συγκρούσεων, χωρίς να το γνωρίζω πολλές φορές. Θεωρούσαμε ότι ήταν ασφαλείς οι περιοχές αυτές και τώρα με την ε, πρόοδο της τεχνολογίας και το ότι έχουν φτάσει τα όπλα και σε κακόβουλα χέρια, δυστυχώς τέτοιες απειλές ε, πολλαπλασιάζονται. Και αυτό θα πρέπει, όπως είπατε, και οι μυστικές υπηρεσίες να ανοίξουν τα χαρτιά τους, να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και αν κάποιες ε, χώρες δημοσιεύουν προειδοποιήσει ε, και απαγορεύουν τι αερογραμμές του να κάνουν υπερτήσει από συγκεκριμένες ζώνες, γιατί να μην το κάνουν και άλλες χώρε. Εγώ ήμουν αεροσυνοδό στην British ε, Airways ε, και πολλές Αεροπορικέ εταιρείε, όπως η Μαλαισία και εκείνη τη μέρα ε, περνούσαν ε, από την ίδια διδρομή. Είχαν την ίδια πορεία πτήση με το Μαλαισιανό. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι ισχύει η θεωρία της συνωμοσία. Επίσης ε, θα ήθελα να πω ότι τα σχέδια της ΕΑΣΑ Κυριακή είναι περιεκτικά και πλήρη. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο ευρωπαϊκό το θέμα. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο γιατί οι φίλοι και οι, οι συγγενείς εργάζονται σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να υπάρχει ένας σωστός και κατάλληλος τρόπος ανταλλαγή πληροφοριών. Να μην απομονωθούμε και να μην οφαλοσκοπούμε και να λέμε ότι εμείς αποφασίσουμε τι θα συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση, γιατί ε, δεν είναι σωστός ο εθνικός τρόπος προσέγγιση, Θα πρέπει να υπάρχει ένα και ο διεθνής τρόπος χαιρετήσω τα βήματά σας ε, και τις προσπάθειές σας ε, και επενώ ε, τις ερευνητικές προσπάθειες. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν και στο μέλλον αυτά τα σχέδια και ε, εγώ έχω εμπιστοσύνη και αύριο θα έμπαινα σε αεροπλάνο και θεωρώ και έχω εμπιστοσύνη και στις μυστικέ υπηρεσίες και στα κρατη Πιστεύω ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και τέλος, ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, αν υπάρχει κίνδυνο κάπου στον κόσμο, είναι δύσκολο να γίνει τέτοια ενημέρωση, γιατί μπορεί κανεί να αγοράσει ένα εισιτήριο από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β και να πει Α, θα περάσετε και από μια επικίνδυνη ζώνη. Είναι δύσκολο να το πει κανεί. Θα πρέπει το κοινό να έχει εμπιστοσύνη στι αρχέ ότι θα, θα προβούν στι κατάλληλε αποφάσει και θα κάνουν τι σωστέ κρίσει με τι πληροφορίε πολύτιμε που δίνουν και οι οργανισμοί επαφή άμεσα σε εσά ότι θα κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Βέβαια, έχει τι καλύτερε προθέσει, κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων έχουμε καλά αποτελέσματα. Δυστυχώ ε, δεν είναι αθώο ο κόσμο και υπάρχουν και πολλοί κακόβουλοι. Και είδατε τι έγινε στο Σάρμελ Σέικ. Δεν ξέρουμε τελικά ακόμη ε, τι γίνεται. Αλλά έχουμε και εμεί ε, παρόμοιε περιπτώσει. Είχαμε το Λόκερμπι, για παράδειγμα, την τραγωδία την αεροπορική του Λόκερμπι. Αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κακόβουλη τρομοκρατία όσο μπορούμε και να υποστηρίξουμε τις αεροπορικές μας εταιρείε και τον κλάδο. Και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε εσάς ότι κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. μπορείτε. Αυτά από το ECR. Ο Ματίας Φων Μίλτεμπεργκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Μιούλερ και τον κύριο Κι για την πολύ σαφή παρουσίασή τους. Δύο ερωτήσει έχω να σα θέσω. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την αξιολόγηση του κινδύνου για το δεύτερο επίπεδο των συστάσεων που περιλαμβάνονται στο, στην έρευνα του Σύμβουλου Ερευνών. Αναφέρεται και παραθέτω ότι αν τα κράτη διαθέτουν πληροφορίες που αφορούν τις πολιτικές πτήσεις, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει με δεδομένη ε, διαδικασία να χορηγηθούν στις αεροπορικές εταιρείες και στους εμπλεκόμενους φορείς. Με διαφθαμένο τρόπο και το τονίζω αυτό. Ε, χαίρομαι που η Άζα συμμετέχει στην κατάρτιση και σε ε, συναντήσεις υψηλού επίπεδου όπως αυτή στο Βουκουρέστη, ε, στην αξιολόγηση λοιπόν των κινδύνων που προκύπτουν πάνω, ε, από τις πτήσεις πάνω από περιοχές συγκρούσεων και που προ, προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις σε ό,τι αφορά ε, και μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Θα πρέπει να σας πω ότι κάποια κράτη δείχνουν περιορισμένη προθυμία να αναγνωρίσουν το ρόλο της ΕΑΖΑ. Πώς το αντιμετωπίζετε λοιπόν αυτό, δεδομένου και ότι το Μάρτιο του 2016 θα προβείτε στην δημοσίευση κάποιων συστημάτων και πορισμάτων και πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτή την αναγνώριση της ΕΑΘΑ από τις ευρωπαϊκές χώρες. Και στο πλαίσιο του ΙΚΑΟ τώρα, στο δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω, αναπτύσσεται μία εφαρμογή στο διαδίκτυο προκειμένου με δομημένο, διαρθωμένο τρόπο να μπορούν να δημοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές στους εμπλεκόμενους φορείς. Πώς αξιολογείται λοιπόν και οι δύο τα εργαλεία αυτά, γιατί χτες έριξα μια ματιά στο, στην ιστοσελίδα και πρέπει να σας πω ότι δεν περιλαμβάνονται πολλές πληροφορίες. Και τέλος, στο τρίτο επίπεδο των συστάσεων τη έκθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ολλανδίας αναφέρεται η ευθύνη των αεροπορικών ε, εταιριών. Θεωρώ ότι υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ της επιθυμίας των, των αεροπορικών εταιριών Τη απροθυμίας των εμπορικών εταιριών να αναφέρουν τις διαδρομέ τις διαδρομές πτήσης τους και τις ανάγκες των ε, επιβατών να γνωρίζουν τα στοιχεία αυτά. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταστήσουμε αυτή την υποχρέωση λιγότερο προαιρετική. Και πιστεύετε ότι χρειάζεται σχετική νομοθεσία. Αυτά ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα ήταν τραγικά αυτά τα περιστατικά και δυστυχώς δεν υπάρχει πανάκια, δεν υπάρχει θαυματουργή λύση. Η αποφυγή των υπερπτήσεων ε, στις εμπόλεμες ζώνες ίσως ε, περιορίσει τους κινδύνους, αλλά ποτέ δεν θα είμαστε 100% σίγουροι και ασφαλείς. Και πώς μπορούμε να προλάβουμε τρομοκρατικές επιθέσεις. Ίσως ε, με καλύτερη συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών, αλλά ούτε και εκεί μπορούμε να είμαστε 100% βέβαιοι ότι θα έχουμε ασφάλεια, γιατί ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ασταθής και όλο και περισσότεροι άνθρωποι ε, βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κίνδυνο. Δυστυχώς ε, έχουμε τέτοια φαινόμενα, αλλά αεροπορικός τομέα είναι ο πιο ασφαλή. 30.000 ε, ε, αεροπλάνα καθημερινά υπερίπτονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάχιστα είναι τα δυστυχήματα αεροπορικέ αεροπορικές Και για να αποτρέψουμε τρομοκρατικέ ενέργειε, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των μυστικών υπηρεσιών και όλων αυτών των οργανισμών που έχουν τόσο χρήσιμο έργο. Ο ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και του δύο σου για την παρουσίαση του Οι συνάδελφοι νομίζω ότι έχουν αναφέρει πάρα πολλέ ε, σωστέ ερωτήσει. Αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ σε μία ερώτηση. Το θέμα τη ευθύνη. Στην παρούσα φάση την ευθύνη την φέρουν ε, οι μεμονωμένε χώρε. Τι θα γίνει λοιπόν στο μέλλον όταν ε, υπάρξει αυτή η High Level Task Force όταν λοιπόν θα πραγματοποιηθούν αυτές οι ιδέες και οι προτάσεις σας θα έχει αυτή η task force συγκεκριμένη ευθύνη, θα συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη ευθύνη. Πώς ε, λοιπόν θα διαμορφωθεί το θέμα της ευθύνης, γιατί δεν φαντάζομαι ότι τα κράτη-μέλη θα δεχόντουσαν να τους αφαιθεί οποιαδήποτε ευθύνη και οποιαδήποτε ε, αρμοδιότητα. Ο Γιουρνοκόλνης. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη δυστυχώς δεν, θα επαναφέρει στη ζωή τους δυστυχείς επιβάτες ε, της μοιραίας πτήσης, αλλά ο κύριος Μίλλερ δεν αναφέρθηκε εκτενώς ε, στην ευθύνη αυτών που εκτόξευσαν τον πύραυλο. Γιατί πολλά αναφέρθηκαν ε, στο θέμα, για το θέμα αυτό και ξέρουμε ότι το υλικό τους ε, δεν ήταν ε, χειροποίητο ή υλικό που βρέθηκε τυχαία στα χέρια τους, αλλά προερχόταν από ένα συγκεκριμένο κράτος. Κάποια στιγμή εκτοξεύτηκαν κατηγορίες και προς την Ρωσία. Γιατί δεν δώσατε περισσότερη συνέχεια στο θέμα αυτό. Επίσης, με εκπλήσει κάπως η πορεία της συζήτησης, γιατί πιστεύω ότι ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές ή τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις, οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες και στη τελική ανάλυση ο διεθνής, ο διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας θα πρέπει να σηματοδοτούν τις εμπόλεμες ζώνες εκεί που οι ε, εμπλεκόμενες πλευρές έχουν στην, στα χέρια τους πυράβλους που μπορούν να έχουν βέλη και να φτάνουν και αεροπλάνα. Δεν μπορούμε να έχουμε στον κόσμο αυτό ε, αντιμαχόμενες πλευρές ε, που να έχουν στη διάθεσή τους τέτοια όπλα και να το αγνοούμε. Θα πρέπει συστηματικά να αποφεύγουμε τις εμπόλεμες αυτές ζώνες σε περίπτωση που έχουν τέτοιες δυνατότητες οι αντιμαχόμενες πλευρές. Νομίζω ότι η κοινή λογική επιτάσσει τέτοιες σκέψεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση και έχω και εγώ κάποιε ερωτήσει να κάνω. Η Task Force η οποία αναφέρθηκε. Στη Γερμανία ξέρετε τι λέμε. Ότι άμα δεν ξέρει τι να κάνει στο μέλλον, ε, φτιάξε εκεί πέρα μια Task Force. Ποιε ε, είναι οι συνέπειε, ποιοι είναι οι όροι συνεργασία όμω, σε ό,τι αφορά το European Single Skies ε, εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε εδώ και ε, πολύ καιρό. Καταρτίζουμε συστάσεις, αλλά παρόλα αυτά μερικέ χώρε δεν τις ακολουθούν τι συστάσεις αυτέ γιατί έχουν πολλού εθνικού εγωισμού και αυτό πάντα ισχύει. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει 100% ασφάλεια, αλλά εδώ δεν γίνεται τίποτα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από από το δυστύχημα τώρα θα προκληθεί μια μεγαλύτερη πίεση στο ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να μπει λίγο ένα όριο στους εθνικούς οργανισμούς και να υπάρξει μια κίνηση. Δεύτερο σημείο. Είπατε ότι μέχρι και την ίδια την ημέρα όλες οι αεροπορικές σχεδόν εταιρείε πετούσαν στον ένα όριο χώρο. Εγώ θυμάμαι ότι διάβαζα σε κάποιες εφημερίδες και πριν το δυστύχημα ότι κάποιες αεροπορικές εταιρείε δεν περνούσαν από τον ενέργειο χώρο αυτό. Ήταν η Λουφτχάνζα. Ποιε ήταν αυτές. Και τέλος το θέμα τη ευθύνη συνδέεται και με την ενοχή, με την ε, υπετιότητα και ξέρουμε ότι υπάρχει δυνατότητα, α, υπήρξε δυνατότητα να συσταθεί στον ΟΗΕ ειδικό δικαστήριο 11 χώρες λοιπόν στις 29 Ιουλίου 2015 ψήφισαν υπέρ της σύστασης τέτοιου δικαστηρίου του ΟΗΕ. Η Ρωσία έφεσε βέτο, αλλά η Ρωσία παρόλα αυτά διατηνόταν ότι δεν φέρει μερίδα της ευθύνης. Σε ό,τι αφορά όμως τον πύραυλο Μπουκ, ήταν από τη Ρωσία, από την Ανατολική Ουκρανία ήταν της Ουκρανίας, Ουκρανικής, ε, των Ουκρανικών αρχών, γιατί και αυτή η κατηγορία ακούστηκε ότι ήθελαν να αμαυρώσουν την εικόνα της Ρωσίας. Ήταν των αποσχιστών. Ασχολείστε με τέτοια θέματα. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω. Έχετε το λόγο. Ε, ehm, Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ερωτήσεις αυτές που θέσατε και τα καλά σας λόγια για την έρευνά μας. Πολλά ε, είναι τα ερωτήματα τα οποία συμπίπτουν. Ε, ο κ. Βαντεκάμπ μας ρώτησε αν υπήρχαν προειδοποιητικέ ενδείξεις. Δεν υπήρχαν προειδοποιητικές ενδείξεις, δεν μας προειδοποίησε ούτε η Eurocontrol όχι τουλάχιστον ρητά. Δεν είναι και καθήκον τους, ούτε κάποια άλλη χώρα. Το μοναδικό το οποίο κάποιοι είχαν κοιτάξει πιο επισταμένως είναι η κατάσταση στην Κρυμαία. Η Κρυμαία είναι λίγο πιο νότια από την Ανατολική Ουκρανία. Η κατάσταση λοιπόν στην Κρυμαία ήταν ε, κάπως ανησυχητική και οδήγησε σε κάποιες αεροπορικές εταιρείες να πάρουμε την απόφαση να επιλέξουν άλλες πτήσεις, άλλες δρομές πτήσεων. Κάποιοι από εσά με ρωτήσατε τι γίνεται, ποιοι πετούσαν πού στις 17 Ιουλίου 2014 και εμείς είδαμε και διαβάσαμε στον τύπο ότι διάφορες εταιρείε δήλωναν ότι δεν πετούν στον αέριο χώρο. Ρωτήσαμε και ζητήσαμε στοιχεία από τη Eurocontrol και ρωτήσαμε λοιπόν ποιοι πετούσαν εκεί. Όλα αυτά περιλαμβάνονται λοιπόν στην έκθεσή μας. Και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι ουσιαστικά όλοι πετούσαν εκεί. Μια-δυο ήταν οι αεροπορικές, οι οποίες για άλλους λόγους δεν περνούσαν από εκεί. Αλλά κανείς δεν απέφευγε τον αερίο αυτό χώρο, συγκεκριμένα λόγω απειλών στην ε, Ανατολική Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε στην έκθεσή μας. Ο κύριος Φαντεν Κάμπ επίσης ε, μας έθεσε και μία ερώτηση για τα δεδομένα των ραντάρ, τα στοιχεία των ραντάρ. Πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό και διαπιστώνουμε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δήλωσε ότι τα πρωτεύοντα δεδομένα του ραντάρ δεν τα είχε. Σύμφωνα με το παράδειγμα 11 τη σύμβαση του ΙΚΑΟ υποχρεούνται να φυλάσσουν τα στοιχεία αυτά, δεν το έκαναν. Γίνεται αναφορά στην έκθεσή μας και φυσικά η έκθεση αυτή διαβιβάστηκε και προς τον ΙΚΑΟ. Δεν υποβάλαμε επίσημα ένσταση, αλλά μπήκε στην ατζέντα του ΙΚΑΟ. Και την προηγούμενη εβδομάδα ένας συνάδελφός μου μετέβησε στο Συμβούλιο του ΙΚΑΟ και το τόνισε και το ανέλησε το θέμα αυτό εκ νέου. Το θέμα για την λίστα των αεροπορικών εταιρείων νομίζω ότι το κάλυψα. Ύστερα, Ρωτήσατε κάποιοι από εσάς το θέμα της κυριαρχίας των κρατών σε ό,τι αφορά ε, τον εναέριο χώρο και ενδεχόμενο κίνδυνο. Είναι δύσκολο και μεγάλο αυτό το δίλημα. Η συνθήκη του Σικάγο έχει ως βάση την κυριαρχία των ε, κρατών. Για να αρθεί αυτή η επικυριαρχία θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, γιατί θα είχε πάρα πολύ μεγάλε συνέπειε, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά για πάρα πολλά ζητήματα. Και δεν το επιλέξαμε λοιπόν αυτό ω οδό. Εμεί ω ε, Συμβούλιο Ασφαλεία είπαμε μόνο ότι το μόνο που μπορεί να ζητηθεί και το μόνο που μπορεί να είναι δυνατόν είναι μια μορφή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, μια ομάδα κρατών αεροπορικών εταιριών, μυστικών υπηρεσιών και ε, οργανώσεων πολιτών. Και εδώ θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σημείο το οποίο το αναφέρατε κι εσείς, ορισμένοι εξημών. Το ερώτημα του κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να δημοσιεύουν στοιχεία και να έχουν ευθύνη για τις πτήσεις τους οι αεροπορικές εταιρείες. Ένας τρόπος λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί προκειμένου εμείς ως επιβάτες να γνωρίζουμε τη διαδρομή της πτήσης και να ξέρουμε ποιοι είναι και οι κίνδυνοι ή πώς έχει γίνει η αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων και φυσικά θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους τους αρμόδιους φορείς, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορούσε και αυτό να αποτελεί ένα μοχλό πίεσης προκειμένου οι αεροπορικές εταιρείες να σκέφτονται πιο καλά τους κινδύνους τους οποίους διατρέχουν αυτό που ανέφερε και η κυρία Φώστερ. Γνωρίζω τον αεροπορικό κλάδο και εγώ επαρκώς και είμαι σίγουρος ότι θέλουν να αντλήσουν τα διδάγματα από τα όσα έχουν συμβεί. Και όπως είπατε και εγώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μπω στο αεροπλάνο γιατί ποτέ πριν δεν ήταν τόσο ασφαλεί οι αεροπορικέ πτήσει στο παρελθόν. Η ΑΖΑ, ο ΙΚΑΟ βλέποντας τι κάνουν όλες αυτές οι εργανώσεις για να περιορίσουν τους κινδύνους διαπιστώνουμε ότι είναι ένας κατεξοχήν τομέας όπου μπορούμε να διδαχτούμε από τα παθήματα του παρελθόντος και νομίζω ότι αυτό το παρουσίασε και επαρκώς και ο κύριος Κι στην παρουσίασή του. Πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, α ναι, μία ερώτηση ακόμα για το από πού προήλθε ο πύραυλος. Εμείς ε, αναφέραμε αναφέραμε ότι προέρχεται από μια περιοχή 340 τετραγωνικών χιλιόμετρων που ήταν στην υπό τον έλεγχο των αποσχιστών, εκεί τερματίζονται τα, τα, μας οι ποινικέ διώξεις ενδεχομένω για την ευθύνη των υπετίων. Είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς δεν, ως Συμβούλιο Ασφαλείας δεν επικεντρωνόμαστε σε θέματα τέτοια ποινική ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση επιπλέον έχει να κάνει ο κύριος Ερτούγκ. Να ρωτήσω τον κύριο Μιούλερ. Η British Airways πριν την κατάρρευση του, της MH17 ήξερε τον κίνδυνο και άλλαξε τις διαδρομές Η απάντηση δεν μπορούμε να επισέλθουμε στα δεδομένα που είχαν οι μεμονωμένες αεροπορικές εταιρείες. Υπάρχουν και τα εμπιστευτικά και τα απόρριτα στοιχεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να σας απαντήσω ότι υπήρχε μία εταιρεία η οποία άλλαξε τι διαδρομέ πτήση. Μπορείτε να πείτε και το όνομα, λέει ο πρόεδρος. Όχι, όχι, δεν επιτρέπεται. Μάλιστα, αλλά είναι σαφές από την έκφρασή σα ποια εταιρεία είναι αυτή. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. έγιναν ε, αρκετές ερωτήσεις για το ρόλο της, του Διεθνούς Οργανισμού ε, της Πολιτικής Αεροπορίας και τον έλεγχο του θέματος. Ο ρόλος, ε, ο κόσμος της πολιτικής αεροπορίας ε, είναι ένας κόσμος που τις περισσότερες αποφάσεις λαμβάνουν τα κράτη-μέλη, τα κράτη. Και τα κράτη είναι κυρίαρχα και τα κράτη-μέλη του ΙΚΑΟ. Οι αποφάσει λαμβάνονται με ομοφωνία. Δεν μπορεί η ΙΚΑΟ να επιβάλλει σε ένα κράτο κάτι που το κράτο δεν θέλει να εφαρμόσει. Και αυτά είναι και τα όρια των εργαλείων που θεσπίζει η ΙΚΑΟ και που στηρίζεται κυρίως σε πληροφορίες για τι προειδοποίησεις γίνονται για απογορεύσεις υπερπτήσεων αλλά δεν μπορείτε να βρείτε εκεί πληροφορίες που προέρχονται από κάποιο κράτος για τον κίνδυνο που ισχύει σε κράτος. Για παράδειγμα το Πακιστάν. Στις αρχές του έτους οι γαλλικές αρχές και κατόπιν οι βρετανικές αρχές δημοσίευσαν ε, σημειώματα για κάποιο κίνδυνο που έχουν οι χαμηλές πτήσεις στο Πακιστάν και ενημέρωσαν αντίστοιχα τις αερογραμμές τους για το κίνδυνο αυτό. Το Πακιστάν ε, διαφωνούσε ριζικά με την εκτίμηση αυτή, γιατί για τις αρχές του Πακιστάν ο κίνδυνος ήταν ιδιαίτερα μικρός. Οπότε ένας διεθνής οργανισμός σαν το ΕΚΑΟ δεν μπορεί να προχωρήσει, να, να πει κάτι στην περίπτωση αυτή. Γιατί Eurocontrol, για πολύ διαφορετικούς λόγους, ε, ξανανοίξαμε ένα τμήμα του αέριου χώρου πάνω από την Κρυμαία που δεν θεωρείται ως ε, εμπόλεμη ζώνη. Και η Ουκρανία ήταν μέρος της Eurocontrol ε, όταν και είπε ότι ξανανοίγω τον αέριο χώρο πάνω από ένα τμήμα της Κρυμαίας. Ήταν δικός ο αέριος χώρος, οπότε η Eurocontrol υποχρεωμένη να ξανανοίξει αυτόν τον αέριο χώρο. Ενώ ναι, εμεί θα πρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση του κινδύνου για να εξετάσουμε την ασφάλεια. Η σύστασή μα ήταν να μην χρησιμοποιηθεί αυτό ο αέριο χώρο πάνω από την Κρυμαία. Αυτά λοιπόν είναι τα όρια του διακυβερνη... των διακυβερνητικών οργανισμών που... στου οποίου ισχύει η ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών και τέτοιου είδου διεθνεί οργανισμοί δεν μπορούν να επιβάλλουν τίποτα στα μέλη του. Τώρα, τι γίνεται στην ε, Task Force υψηλού επίπεδου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα και δεν είναι σίγουρα η βέλτιστη λύση. Ελπίζω να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα αυτή την task force και να πολλαπλασιάσουμε τις επιμέρους ομάδες. Αλλά αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε αυτή την ομάδα κρούση, αυτή την task force, γιατί είχαμε ε, κολλήσει σε διέξοδο. Γιατί όλοι συμφωνούσαμε ότι υπάρχει καθήκον για ανταλλαγή πληροφοριών. Κανένα, ούτε στι μυστικέ υπηρεσίε, ούτε στι στρατιωτικέ αρχέ, ούτε στι εθνικέ διοικήσει ε, δεν θα έλεγε αρνούμε να ανταλλάξουμε πληροφορίε για την ύπαρξη συγκεκριμένου κινδύνου. Δυστυχώ όμως ε, και εκεί και τη δυσκολία κάποιες χώρες που έχουν στρε... Ε, ανεπτυγμένες υπηρεσίες και πολλές πληροφορίε, πληροφορίες ενώ άλλε ε, περισσότερες χώρες μέλη δεν έχουν τέτοιες πληροφορίε και ζητούν ευρωπαϊκή διαδικασία για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις στρατιωτικές πληροφορίες που έχουν λίγες μόνο χώρε. Και εκεί είναι που κολλήσαμε. Γιατί έχουμε δύο, τρει, τέσσερι χώρε που λένε εμεί δεν χρειαζόμαστε την Ευρώπη, γιατί έχουμε τι δικέ μα πληροφορίε, ενώ οι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε λένε θέλουμε την Ευρώπη, θέλουμε ευρωπαϊκή λύση για να έχουμε πρόσβαση σε αυτέ τι πληροφορίε. Αυτό το γόρδιο δεσμό προσπαθεί να λύσει αυτή η ομάδα δράση ε, και τη συστήσαμε για να μπορέσουμε να έχουμε ήδη αποτελέσματα πολύ γρήγορα και στη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας και μάλιστα ε, σας καλούμε, είναι ανοιχτή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η Task Force, θα συνεδριάσει τρεις φορές και θα πρέπει το Μάρτιο ήδη να αποφέρει καρπούς. Αν δεν ε, είναι αποδοτική μέχρι το Μάρτιο θα διαλυθεί αυτή η Task Force. Οπότε υπάρχει ηθικό καθήκον όλων και όλοι το αντιλαμβάνονται. Έχουμε κολλήσει λίγο στους τρόπους και στη μεθοδολογία. Πώς θα, ε, θα συγκεντρώσουμε αυτές τις πληροφορίες και πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό θα είναι το επόμενο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε. Γιατί με κάποιες χώρε έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Γιατί λένε οι χώρες αυτές ότι το μόνο σώμα που μπορεί να έχει πρόσβαση στις εθνικές τους αερογραμμές είναι οι εθνικές αρχές και όχι οι ευρωπαϊκές αρχές η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι με την ευρωπαϊκή ενία αγορά, με τους κοινούς κώδικες, με τις ε, συμμαχίες, με τις, τους, τις ομάδες των οργανωτών, δεν είναι δυνατόν ε, να έχουμε τέτοια στεγανά συστήματα. Γιατί πολλοί επιβάτες που παίρνουν, Γάλλοι που παίρνουν την KLM δεν γνωρίζουν για τις πληροφορίες που ε, αντιμετωπίζουν, που ανταλλάσσουν οι Ολλανδικές με τις ε, Γαλλικές αρχές. Συνήθως είναι κοινέ ε, αυτές οι πτήσεις. Και επίσης ε, για τους τρομοκράτες δεν έχουν όλε οι πτήσει την ίδια αξία. Οι τρομοκράτε προτιμούν να χτυπήσουν ένα βρετανικό, ένα γερμανικό αεροσκάφο, ένα αμερικανικό ή ένα ρωσικό, εν προκειμένου. Γιατί η πολιτική αξία και ο πολιτικό συμβολισμό είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό ισχύει. Και εκεί έγκυται και μία από τις δυσκολίες, ότι δεν ισχύει ο ίδιος κίνδυνος για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Αλλά σε τελική ανάλυση, οι πολίτες πετούν με ευρωπαϊκές ή μη ευρωπαϊκές αεροπορικές γραμμές ε, και θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι όλες αυτές οι αεροπορικές εταιρείε έχουν τις ε, πληροφορίες που χρειάζονται για να πραγματοποιούν ασφαλείς πτήσεις. Αυτή είναι η δυσκολία μας όμως. Προσπαθούμε με αυτή την Task Force να σημειώσουμε πρόοδο και εκεί έχουμε κάποιες χώρες μέλη μερικές που έχουν τις πληροφορίες που είναι οι ε, κύριοι των πληροφοριών και άλλοι που είναι αποδέκτες των πληροφοριών προσπαθούμε να συμβιβάσουμε τα διάφορα συμφέροντα και να επικρατήσει η κοινή λογική στον τρόπο ανταλλαγής των πληροφοριών. Πάντως, <laughs> το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις δύο πολύ ενδιαφέρουσες αυτές παρουσιάσεις και για τη συζήτηση αυτή που κάναμε και για τις ερωταπαντήσεις λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ασφαλώς και δεχόμαστε με μεγάλη ευχαρίστηση ε, την ε, πρόθεση να μας αναφέρει τα προς τα απορίσματά της. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε λοιπόν ε, στις 3 το απόγευμα για την ακρόαση.